So, dear colleagues, please uh, take a seat so that... Καθίστε παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε.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 Ο πρόεδρος λέει ότι οι διερμηνείς θα κάνουν ένα μήνυμα, Dispute. θα κάνουν μια ανακοίνωση για την εργασιακή τους διένεξη και την κατάσταση που επικρατεί στην υπηρεσία τους. Θα επαναλάβουμε λοιπόν ε, το μήνυμα αυτό οποίο είπαμε και στην αρχή, πω βρισκόμαστε στην τρίτη εβδομάδα κινητοποιήσεων λόγω τη εργασιακή διένεξη με τη διοίκηση, λόγω τη επιστράτευση ορισμένων καμπινών που καταργεί το δικαίωμά του στην απεργία και συνιστά διάκριση και προ τι υπόλοιπε γλώσσε, ένδειξη αλληλεγγύη η ελληνική καμπίνα σήμερα δεν θα προχωρήσει στην προβλεπόμενη στάση εργασία. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία και νομίζω ότι όλοι μας ε, θέλουμε να βρεθεί μια ικανοποιητική για όλους λύση. Μας ενδιαφέρει να λυθεί αυτή η διένεξη ώστε να μπορέσουν οι διεμείς να συνεχίσουν ε, το έργο τους και να υπάρχουν ε, και οι σωστές σχέσεις εδώ στο Κοινοβουλίο. Ερχόμαστε στη Μελισσιαδιάταξη. Υπάρχει κάποια πρόταση, όχι, άρα εγκρίνεται η μεσιάδεξη. Δεύτερο σημείο της μεσιάς διάταξης, έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων. Ως συνήθως ε, τα πρακτικά θα θεωρηθούν εγκεκριμένα εάν δεν έχουμε κάποια παρατήρηση μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Και σημείο 3, ανακοινώσεις ε, σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών. Και στην περίπτωση αυτή αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, θα θεωρηθεί ότι εγκρίνονται οι αποφάσεις των συντονιστών. Σημείο 4. Ανακοινώσεις της Προεδρίας. Να πω ότι ως συνήθως μεταδίδεται στο διαδίκτυο η συνεδρίασή μας από την ε, Νιρεμβέργη μέχρι το Γκέτεμπορκ ε, και μέχρι την Λουμπλιάνα. Θέλω να καλωσορίσω όλους όσους μας ακούν. Υπάρχει διερμηνία επίσης. Ε, μπορείτε λοιπόν να μιλάτε αργά καθαρά και έτσι θα μπορέσουμε να ε, ακούσουμε ξεκάθαρα τα μηνύματα που θέλετε να μεταφέρετε. Σημείο 5. Είναι μαζί μας ε, ο Γενικός Διευθυντής ε, της ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Εμπόριο, DigiTrade, ο Ζαν Λουκ Ντεμαρτή, τον οποίο καλωσορίζουμε. Θα μιλήσουμε μαζί του για τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΑ, ιδίως μετά την επιβολή δασμών στο χάλιβα, το αλουμίνιο και τις αποφάσεις τις σχετικές. Είχα μετά την απόφαση του Τραμπ προβεί σε μια δήλωση ε, λέγοντας ότι είναι σαφές πως καταδικάζουμε την απόφαση αυτή που θεωρούμε και ότι είναι παράνομη σε ό,τι αφορά τους κανόνες του ΠΟΕ. Στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή την προσέγγιση ε, τριών ε, σταδίων που έχει υιοθετήσει και νομίζω ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ομοψυχία και την ενωμένη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελπίζοντας να παραμείνουμε ενωμένοι στη συνέχεια. Και τώρα, βεβαίως, μετά την απόφαση για το χάντουβα και το αλουμίνιο ε, προσθέθηκαν και άλλα. Ε, είχαμε την ανακοίνωση ότι θα υπάρξει έρευνα για την επιβολή πρόσθετων δασμών στα αυτοκίνητα. 2-3-2. Ε, εθνική ασφάλεια, αυτό ήταν το, η νομική βάση για τον πρόεδρο Τραμπ. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως. Όσο πια ε, τα αυτοκίνητα μπορούν να βλάψουν την εθνική ασφάλεια των Αμερικανών. Καλό θα ήταν να ακούσουμε κάποιες διευκρινήσεις. Ε, ξέρετε τι έγινε και στη, στη γενική, στην συνάντηση της ομάδας των 7 μετά από τρεις ημέρες Statement related to these uh, duties, which is um, Ανακοινώθηκε ότι θα επιβληθούν και στην Ισπανία δασμοί για τις ελιές. Άρα βλέπουμε πραγματικά ε, ένα ντάμπινγκ και μια επίθεση κατά της κοινή γεωργικής πολιτικής. Πολλά είναι τα ζητήματα και πολλές οι απορίες που έχουν γεννηθεί. Ζανλίκ, τι απαντήσεις να μας δώσεις εσύ. Ευχαριστώ πολύ, Μπέρντ. Ναι, πράγματι. Δύσκολη καιροί που ξεκινούν στις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πολλές δυσκολίες. Όχι μόνο διμερός, αλλά και στο πλαίσιο του παγκόσμιου εμπορίου και της παγκόσμιας οικονομίας. Πραγματικά είναι πολλές οι προκλήσεις ε, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε διάφορα μέτωπα. Τις ε, τελευταίους μήνες ε, είδαμε να επιβάλλονται στο τμήμα 232 δασμοί βάση υποτίθεται ανησυχιών για την εθνική ασφάλεια από ψυχροπολεμικές εποχές. 2-3-2 λοιπόν, δασμοί στο αλουμίνιο και στο χάλιβα. για τη Ρωσία και το Ιράν έχουμε κυρώσει. έχουμε μια νέα εθνική έρευνα στην Αμερική. Ένα ε, πρόβλημα επίσης ε, στη, στο πλαίσιο του ΠΟΕ και στην ε, σύνοδο του G7 επίσης ε, ήταν αρνητικές εξελίξεις. Και άλλοι δασμοί πρόσφατα δυσανάλογοι στους ελιές, στις πανικές. Αναλύουμε την κατάσταση και είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας στο πλαίσιο πολυμερούς εμπορικού συστήματος. Αυτοί οι δασμοί 232 για το χάλιβα και το αλουμίνιο επηρεάζουν και δημιουργούν μεγάλη ζημία by the US domestic industry. Δεν είναι κατάλληλο μέτρο η προστασία ενός ολόκληρου τομέα αν υπάρχει πρόβλημα υπερλεονάζοντος δυναμικού, πλεονάζοντας παραγωγής. Δεν λύνεται αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να υπάρχει αναλογία, ανάλογες απαντήσεις, όχι τις ανάλογες. Ξεκινήσουν νομικές διαδικασίες στο πλαίσιο του ΠΟΕ και μάλιστα ήδη ξεκίνησαν οι διαδικασίε οι δεσμοι 2 δασμοί 2-3-2 και την προηγούμενη Πέμπτη όλα τα κράτη συμφώνησαν να προχωρήσουν με μια επανεξισορρόπηση. Θα ασκήσουμε δηλαδή τα δικαιώματα εξορρόπησης μέχρι του ε, του 2,8 δις εξαγωγών τις επόμενες ημέρες. Άρα ο κανονισμός που επιβάλλει δασμούς σε ορισμένα προϊόντα θα δημοσιοποιηθεί στην επίσημη εφημερίδα πολύ σύντομα και θα αρχίσουν να ισχύουν την επομένη της δημοσίευσής τους. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε την ενωσιακή αγορά από τις τρέβλες αγοράς λόγω κλεισίματος της αγοράς των ΗΠΑ. Πρέπει να αντιδράσουμε στέναρα και με ομοψυχία γιατί έτσι θα στείλουμε ένα σαφές μήνυμα της δυνατότητας και της ε, ικανότητας που έχουμε να αντιδράσουμε ενωμένοι. Είμαστε ενωμένοι ε, και σε ό,τι αφορά τη νέα έρευνα εθνικής ασφάλειας ε, για τα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά τους, τα εξαρτήματα. Ό,τι εξέλιξη έχουμε στην αυτοκίνητο βιομηχανία θα επηρεάσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την παγκόσμια οικονομία εν γέννη. Αλλά και την Αμερικανική οικονομία. Τέτοια μέτρα θα έχουν επίπτωση και στην Αμερικανική οικονομία. Πιο σημαντικά θα είναι δε και πιο αρνητικά για τη ΣΥΠΑ από ό,τι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι άλλοι εμπορικοί εταίροι θα προβούν σε αντιμετρά. θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διαχειριστούμε στον εδώ καλύτερα αυτή την κατάσταση, αλλά φυσικά ε, όλα αυτά δημιουργούν ένα μεγαλύτερο κλίμα αβεβαιότητας και είναι λυπηρό ε, που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τώρα και τις συστημικές επιπτώσεις αυτών των ε, πολιτικών και για το πολυμερές εμπορικό σύστημα. Ο πρώτος Τραμπ Δεν φαίνεται να έχει διαβάσει τον Ρικάρντο, τον Άνταμ Σμιθ και άλλους μεγάλους οικονομολόγους και το βλέπουμε και από την απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου τη προηγούμενη εβδομάδα που επιβάλλει δυσανάλογε απαγορομετευτικού δασμού ε, ε, στι ελιέ ε, από την Ισπανία. Ήδη η Ισπανία έχει μεγάλη απώλειες στις εξαγωγές της. Είναι μεγάλο πλήγμα για τους αλληλοπαραγωγούς της Ισπανίας που είναι η βασική πηγή εισοδήματός τους οι εξαγωγές αυτές. Είναι σαφές ότι μπορούμε μόνο το χειρότερο να περιμένουμε μετά από όλα αυτά. Πέραν της οικονομικής δυσκολίας και δυσχέρειας των Ισπανών ελοπαραγών που θα πληγούν, θεωρούμε ότι θα υπάρχουν συστημικές συνέπειες από αυτή την απόφαση και αυτό που ζητούμε είναι να μην ανοίξει το κουτί της Πανδώρας για τους ε, Δεν εισακούστηκαν οι κλήσεις μας όμως. Υπάρχει ε, ο Οργανισμός Προστήξης Προϊόντων Επίσης, εθαμό, αμύγδαλα, αραβόσιτος και άλλα προϊόντα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά δεν είναι στο πράσινο κουτί, ε, όπως άλλα προϊόντα στο πλαίσιο των ε, διαβλέσεων με τις χώρες ΑΚΕ. Και όλα αυτά θα, θα τα δούμε. Για να δούμε τι πρέπει να γίνει σε επίπεδο στήριξης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα ισχυρό εμπορικό σύστημα. Πρέπει να σκεφτεί πώς θα το εξυγχρονίσει το σύστημα αυτό να είναι κατάλληλο για τον 21ο αιώνα, προσαρμοσμένο στις νέες ανάγκες. Θα πρέπει όμως να διαχειριστούμε ταυτόχρονα τις διατλατικέ σχέσεις, κατά τρόπον που να προκύψουν ώστε το λιγότερες ζημίες για την παγκοσμία οικονομία. Αυτό σημαίνει πρώτον να είμαστε σταθεροί, στεναροί απέναντι στη ΣΥΠΑ όταν αυτό χρειάζεται, αλλά και να είμαστε αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε και χώρες όπως η Κίνα, που έχει μεγάλη ευθύνη πρέπει να καταργήσει τις ε, διακριτικές εμπορικές τις πολιτικές και να βοηθήσει να υπάρξει αποκατάσταση εμπιστοσύνης. Υπάρχει δρόμος, μπορούμε με τριγωνικό τρόπο, Ευρωπαϊκή Ένωση, Κίνα, είπα να, το τρίγωνο αυτό δηλαδή, να δώσουμε το καλό παράδειγμα για χώρες απέναντι, μάλλον όπως είναι η Ιαπωνία, ο Καναδάς, το Μεξικό, Κορέα, η Αυστραλία. Δεν είναι εύκολο, αλλά θα το προσπαθήσω. Τέλος, θέλω να σας ευχαριστήσω για την ειλικρινή σας υποστήριξη. Διαστόματος του Προέδρου σας. Είπατε ότι στηρίζετε την προσέγγιση Κομισιόν μέχρι τώρα. Οι επαφές σας με το Κογκρέσο είναι σημαντικές. Ε, έχουμε τις μεσοπρόθεσμες εκλογές, σύντομες είπα και παρακαλώ να μεταφέρετε στους ομολόγους σας από τη ΣΥΠΑ τις ανησυχίες μας για την εμπορική πολιτική. Στη Γερουσία, στο Κογκρέσο, οι ομολογοί σας έχουν τη δύναμη να προσπαθήσουν να αναστρέψουν ε, την κατάσταση και να αποφύγουμε χειρότερα όπως αυτό για τα αυτοκίνητα και τα εξαρτήματα ε, των ε, οχημάτων που θα ήταν καταστροφικά για την οικονομία. Any Σας ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν παρατηρήσεις ή ερωτήσεις. Δεις. Ε, Ρούμπικ. Ο κύριος Ρούμπικ. Η ερωτησεις ρουμπικ ο κυριος εχει το λόγο. Ευχαριστώ. Αναφερθήκατε στο rebalancing και το γεγονός ότι θα λάβει η χώρα με βάση τους κανόνες ε, ε, του ΠΟΕ. Και πώς θεωρείτε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο επίπεδο του δευτεροβάθμιου ιδιωτικού όργανου του Appellate Body. Ε, μήπως εκεί θα περιοριστούν αρκετά οι δυνατότητες που έχουμε λοιπόν. Μήπως για παράδειγμα σε επίπεδο ΠΟΕ θα είχαμε τη δυνατότητα σε πολυμερές επίπεδο να αναλογιστούμε το κατά πόσο θα μπορούσε να δοθεί μια συνέχεια σε αυτό το Appellate Body και πολυμερός. Ευχαριστώ. Συμφωνώ ε, με αυτά που είπε ο πρόεδρος Λάγκη ότι στηρίζουμε την πολιτική της Κομισιόν. Έχω δύο συγκεκριμένα ερωτήματα όμως. Σε ό,τι αφορά επιτραπέζιες ελιές, είπατε ότι δεν θέλετε να ανοίξει το κουτί της Πανδώρας. Πώς όμως ε, θα αντιδράσουμε με αποφασιστικά, ισορροπημένα και προσεκτικά μέτρα για την κατάσταση αυτή που έχει δημιουργηθεί και η οποία φυσικά δεν επηρεάζει μόνο τις ε, σπανικές ελιές αλλά μπορεί να θέσει σε κίνδυνο και την κοινή γεωργική πολιτική. Ε, φαντάζομαι ότι είναι μέσα στα μέτρα που εγκρίνονται στο ΠΕΣ Είπατε ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξαναδεί τις σχέσεις της με τους υπόλοιπους εταίρους και να ε, καθορίσει η συντονισμένη πορεία και δράση, γιατί αυτό θα μας δώσει μεγαλύτερη ισχύ. Συμφωνώ. Πώς όμως βλέπετε τις σχέσεις με τη Ρωσία. Πώς μπορεί η σημερινή κατάσταση να επηρεάσει τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορούμε να συζητήσουμε για την σημαντικότατη αυτή πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για μία ακόμα φορά βέβαια. Θα ήθελα να σας πω ότι είχαμε και τη δυνατότητα να συζητήσουμε το ζήτημα αυτό και στο παρελθόν και προφανώς στηρίζουμε, αυτό είναι τις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενωμένοι στεκόμαστε και εμείς και τα κράτη-μέλη. Διάβασα χθε, αν δεν κάνω λάθο, στο Reuters ότι υπάρχουν ήδη κάποιε πρωτοβουλίε που ενδεχομένω να εγκρίνει το Συμβούλιο για τη μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και ξέρετε ότι ε, μία από τις επικρίσεις των ΗΠΑ είναι η εκαζόμενη αποτυχία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Μπορείτε να σχολιάσετε καθόλου τις ε, πρωτοβουλίες αυτής του Συμβουλίου ή μεμονωμένες πρωτοβουλίες των κρατών μελών. Επίσης, θα μπορούσατε να αφαιρθείτε λίγο στις, ε, στην κλιμακούμενη αυτή ένταση μεταξύ των ΗΠΑ και Κίνας και πώς αυτό ενδεχομένως να, παρουσια... να επηρεάσει εμάς στην Ευρώπη και τι παραπάνω θα μπορούσαμε να κάνουμε ως προς αυτό. Ο Κριστόφ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Γενική Διευθυντή, σας ευχαριστώ για τις ε, παρατηρήσεις σας. Ένας ε, καλός μου φίλος ε, μου είπε μια φορά ότι στα πλαίσια εμπορική σύγκρουση και εμπορικού πολέμου μπορούμε να πούμε ότι έχουμε δύο άτομα τα οποία στέκονται το ένα απέναντι από το άλλο, χτυπώντα ουσιαστικά τον εαυτό του και περιμένοντα ότι ο άλλο θα καταρρεύσει πρώτο χωρίς να θέτω να αμφιβόλω σαφώς την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μολονότι είναι σημαντικό να συζητήσουμε και τη δική μας στάση και την αναλύσουμε περισσότερο, αν και θεωρώ ότι είναι εύλογη, θα πρέπει καταρχάς να δούμε τι θέλουμε να πετύχουμε με το rebalancing, την εξισορρόπηση. Ξέρω ότι ο Καναδάς έκανε μία έρευνα προκειμένου να δουν αν τα δικά τους ε, μέτρα εξισορρόπησης, αντιστάθμισης δεν θα επηρέαζαν τους καταναλωτές. Μπορούμε κι εμείς να κάνουμε κάτι το ανάλογο. Είναι πολύ δύσκολο να καταφέρουμε να το εξηγήσουμε αυτό στους Ευρωπαίους πολίτες ή εγώ ας πούμε στους ε, δικούς μου ψηφοφόρους, στους απλούς πολίτες οι οποίοι ε, πηγαίνουν σε σούπερ μάρκετ και θα πρέπει να πληρώνουν πλέον πολύ πιο ακριβή τιμή για να αγοράσουν κάποια αμερικανικά τρόφιμα, φασόλια για παράδειγμα από την Αμερική ή κάτι τέτοιο. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, το ότι μπορεί να υπάρχουν αντίμετρα και πέρα από τα αυτοκίνητα και τα εξαρτήματα αυτοκινήτων. Από ό,τι φαίνεται το αμερικανικό βίσκι το Bourbon είναι στον κατάλογο αυτό. Ξέρουμε ότι τα υνοπνευματώδη ποτά όμως αποτελούν πολύ σημαντικό, παραγωγικό, μάλλον πολύ σημαντικό προϊόν εξαγωγής και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως κλιμακωθεί ένταση και ξαφνικά επιβληθούν δασμοί και στα δικά μας υνοπνευματώδη ποτά. Και μία ερώτηση κάπως φιλοσοφική τώρα. Όταν παραβιάζει κάποιος τον νόμο θα πρέπει να προσάγεται στη δικαιοσύνη. Αυτό γίνεται κανονικά. Και όταν το έθεσα αυτό στην διαχειριστική ομάδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, είπα ότι θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε, μάλλον ποιες είναι επιπτώσεις του να κερδίσουμε ή να χάσουμε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Αν χάσουμε τα πράγματα είναι απλά. Στην πράξη ουσιαστικά θα κριθεί νόμιμη η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών τα μέτρα τους θα θεωρηθούν νόμιμα και θεμητά και ενδεχομένω και άλλες χώρες να ακολουθήσουν το δρόμο των ΗΠΑ και τις δικές τους πρακτικές. Με έχει απασχολήσει όμως πολύ ποιε είναι οι επιπτώσει μια δική μα νίκη στην προσφυγή αυτή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Αν ο ΠΟΕ αποφασίσει τελικά ότι παραβιάζονται οι κανόνες τότε εμείς τι θα κάνουμε. Μπορούμε πραγματικά να σταθούμε στο ύψο των περιστάσεων, να νικήσουμε Πώ θα αντιδράσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πει ο Τραμπ πάρα πολύ ωραία. Ο ΠΟΕ είπε ότι δεν είναι νόμιμα και θεμητά τα μέτρα μέσα, επομένως θα τα σταματήσουμε. πώς ξαφνικά οι Ηνωμένες που είναι πολύ ωραία αποχωρούμε και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Αυτό νομίζω θα πρέπει να μα απασχολήσει. Δεν είναι λάθο αυτό το οποίο κάνουμε, ούτε είναι λάθο η προσέγγιση μα, αλλά θα πρέπει στο πλαίσιο αυτό να δούμε ποιε ήταν οι επιπτώσει και στη μία και στην άλλη πλευρά. Μα θα του στείλουμε την αστυνομία τη Σουηδία. Μα δεν έχουμε, δεν έχουμε, μην ανησυχείτε. Ε, θα αναφερθώ στις τελευταίες παρατηρήσει που έκανε ο κύριο Ευθύνη. Ε, καταρχήν να ευχαριστήσω για την ενημέρωση που ακούσαμε ε, και εγώ συμφωνώ ότι θα πρέπει να προσεγγίσουμε το ζήτημα λίγο ευρύτερα, πέραν δηλαδή των άμεσων εμπορικών κινδύνων που αντιμετωπίζουμε μέσω τέτοιου είδου ακυρώσεων ή μέσω αυτή τη αύξηση των δασμών. οδηγούμενοι δηλαδή μέρα σε μια σύγκρουση στις σχέσεις μας. Νομίζω πως εδώ ο στόχος είναι ο ΠΟΕ και η Κίνα από την πλευρά δηλαδή της πολιτικής ε, που εφαρμόζει αυτή την περίοδο η κυβέρνηση Τραμπ. Οπότε μήπως θα πρέπει να αναλογιστούμε ποια θα πρέπει να είναι η απάντηση, η αντίδραση που θα έχουμε από τη δική μας πλευρά σε πολυμερές επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη και την Κίνα και το ΠΟΕ. Ε, δηλαδή ποια είναι η στρατηγική μας όταν για παράδειγμα ε, έχουμε μια αύξηση των δασμών από την πλευρά των ε, ΗΠΑ απέναντι στην Κίνα, προβαίνουμε και εμείς σε μια αντίστοιχη αίσθηση των δασμών απέναντι στην Κίνα. Θα πρέπει λοιπόν να αναλογιστούμε ποιος, ποια είναι η στρατηγική μας. Ε, και να δούμε ε, ποια είναι η πολιτική της Αμερικής. Αν η Αμερική πραγματικά ε, ακολουθεί το δόγμα του, η Αμερική πρώτα και εμείς θέτουμε τους κανόνες και άλλοι πρέπει να συμμορφώνονται, πράγματι βρισκόμαστε σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Οπότε θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα λάβει η Επιτροπή κατά τον επόμενο μήνα, ούτω ώστε να προβεί σε μια ευαισθητοποίηση, αν θέλετε, των κρατών μελών ως προς αυτό το ζήτημα. Προκειμένου η Επιτροπή να αποκινούμε άλλες χώρες να μιλήσει με, με σαφή και ξεκάθαρη γλώσσα απέναντι στις ε, Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, δηλαδή ε, να πούμε στην Αμερικανική πλευρά ότι δεν σας νοιάζει τελικά δηλαδή η διεθνή θεσμική δομή, δεν σας νοιάζουν οι διεθνείς κανόνες, πράγμα το οποίο δεν μας οδηγεί πουθενά αυτό θα πρέπει να το πούμε, αλλά ε, πείτε μας, ε, κύριε ε, Γενική Διευθυντά, ποια θα είναι τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα λάβουμε μέσα στο επόμενο. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τους δασμούς για το χάλιβα, θα θέσουμε από κοινού τους κανόνες και τους όρους που θα θέσουμε μαζί με τους άλλους. γιατί τα προϊόντα τα οποία ε, τελικά δεν καταλήγουν στην αμερικανική αγορά θα καταλήξουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Οπότε δεν λύνουμε κάτι. Ε, θα πρέπει να βρούμε κοινέ λύσει απέναντι σε αυτό το ε, πρόβλημα. Και ίσως και ο Σά θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πολύ καλό τέτοιο θεσμικό όργανο, μια θεσμική δομή μέσω της οποίας θα μπορούσαμε να συζητήσουμε από κοινού αυτά τα ζητήματα περί επιβολής εντασμών. Ο κύριος Σάνφελτ σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να πω ότι σε περιόδους ε, κρίσης αυτό που ε, παρατηρούμε συχνά είναι ότι όσο πιο άσχημη είναι η κατάσταση τόσο περισσότερες πιθανότητες ε, υπάρχουν για να βελτιωθεί. Οπότε ε, η ερώτησή μου προς τον κύριο Γενικό Διευθυντή είναι η κατάσταση εδώ μπορεί να βελτιωθεί πράγματι ή μπορεί να επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο. Ε, θυμάμαι ότι τον τελευταίο Σεπτέμβριο είχαμε ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα ως προς το ότι δηλαδή αν είχε ξεκινούσε ο εμπορικό ε, πόλεμος ε, θα μπορούσε να ε, περιλάβει μία σειρά από περαιτέρω κλάδους. Οπότε το ερώτημά μου είναι, αυτή η σύγκρουση, αυτή η διαμάχη ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένε Πολιτείες γιατί έτσι την αντιλαμβάνομαι εγώ, ως διαμάχη ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ, όχι ανάμεσα στις ΗΠΑ και το υπόλοιπο κόσμο, μήπως θα πρέπει να μας οδηγήσει ε, σε μία συζήτηση ως προς τις διμερείς σχέσεις, μήπως θα πρέπει να αρχίσουμε δηλαδή να αναλογιζόμαστε πάλι τη συμφωνία τύπου TTIP. Και αυτό το ρωτάω γιατί ε, άκουσα κάποιες... Ε, ε, δηλώσεις ε, τις τελευταίες εβδομάδες, για παράδειγμα πριν από δύο εβδομάδες από τον τον ε, αλλά και από την κατηλάριο Μέρκελ πριν από δύο εβδομάδες. Και σε αυτές τις δηλώσεις του, σε αυτές τις δηλώσεις του αναφέρθηκαν σε ένα είδος μικρής τύπου. Οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχουν κάποιες σκέψεις από την πλευρά της Επιτροπής ε, ως προς αυτό το ενδεχόμενο του να επιστρέψουμε δηλαδή σε ένα διμερές επίπεδο σχέσεων ε, με τις ε, Ηνωμένε Πολιτείε. γιατί ενδεχομένως ε, σε μια τέτοια ευρεία διαπραγμάτευση οριζόντιου χαρακτήρα ε, δεν θα είχαμε πρόβλημα να λύσουμε τα επιμέρους προβλήματα που παρατηρούνται σε ε, μεμονωμένους κλάδους. Για παράδειγμα, στον τομέα του Χάλιβα είναι τόσο άσχημα τα πράγματα ε, έτσι ώστε πραγματικά να μπορούν μόνο να βελτιωθούν ή υπάρχουν περιθώρια να επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Σαλαφράγκα. Ε, Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Ντεμαρτή, στον οποίο έχω κάποιες ερωτήσεις να θέσω. Πρώτη ερώτηση, αν μπορείτε να μας ξαναπείτε ποιος είναι ο ποσοτικός αντίκτυπος των μέτρων ε, στους τομείς χάλιβα και αλουμινίου και αν έχετε υπολογίσει ε, ενδεχόμενα περιοριστικά μέτρα και για τα αυτοκίνητα τι επτός θα είχαν. Δεύτερον, για την G7 και ξέρουμε ότι υπήρξε διαφωνία στο τέλος με τον ανακοινωθέν πού οφείλεται αυτή η διαφωνία και κατά πόσον ε, οι επιπτώσεις ε, της συνάντησης των G7 θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση της συμφωνίας ναύτα. Σε μια στιγμή ιδίω που και θέλω να συγχαρώ την Κομισιόν γι' αυτό, έχουμε ε, ανανεώσει την συμφωνία σύνδεσης με το Μεξικό. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω να εκφράσω την ανησυχία μου και εγώ κύριε Πρόεδρε για το θέμα των Ισπανικών ελιών όχι μόνο για τη βλάβη και τη ζημία για τους παραγωγούς αλλά όπως και ο κύριος Δεμαρτή γιατί αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει προηγούμενο και να επηρεάσει την όλη γεωργική πολιτική, την κοινή γεωργική πολιτική και συμμερίζομαι την υποστήριξη που εξέφρασε ο Πρόεδρος στην Κομισιόν για τα μέτρα που έχει λάβει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Thank you, Director General. Sorry to be delayed this morning. Ο Κάμπελα. Σας ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα, κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να ακολουθήσουμε την ακόλουθη τακτική, δηλαδή να μην προχωρήσουμε σε αντίμετρα και σε αντίπεινα, να επιβάλλουμε δηλαδή και εμεί δασμού, γνωρίζοντα το χαρακτήρα του Ντόναλτ Τραμπ. Αυτό θα είναι μάλλον αντιπαραγωγικό. Και τότε πραγματικά θα καταλήξουμε σε εμπορικό πόλεμο, γιατί αυτό θα απαντήσει στα δικά μα τα αντίπεινα και ούτω καθεξή. Τα δασμολογικά αυτά μέτρα, από ό,τι φαίνεται, μάλλον μπορεί να λειτουργήσουν αρνητικά ακόμα και για τις Ηνωμένε Πολιτείε και να είναι επιζήμια γενικά και για τη δική τους τη χαλιφουργία. Μήπως θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε εμείς μία άλλη τακτική και να αποφύγουμε τελικά τον εμπορικό πόλεμο, γιατί πολύ φοβάμαι ότι αν εμείς θεσπίσουμε κάποια αντίπινα και αντίμετρα, θα απαντήσει με επιπλέον τέτοια αντίμετρα και ο πρόεδρος Τραμπ. Δεν ξέρω λοιπόν αν θα πρέπει να κάνουμε ένα διάβημα μέσω του ε, Λευκού Οίκου ή άλλων θεσμικών οργάνων και να πούμε τελικά ότι τα μέτρα αυτά τα δικά τους είναι μάλλον αυτοκαταστροφικά, εναντίον τους επιστρέφουν. Η κυρία Ρενά έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Δεν είχα την πρόθεση να πάρω το λόγο, αλλά μετά την παρέμβαση του συναδέλφου του ΕΛΚ πραγματικά μου προκαλεί εντύπωση ότι θεωρούν ότι, μπορούμε, ότι μπορούν πραγματικά να συνεργαστούμε διμερώς με τις ΗΠΑ, ενώ οι ΗΠΑ δεν σέβονται τα πολυμερή μέτρα και τους πολυμερείς κανόνες. Νομίζω πραγματικά ότι σε ένα διμερές επίπεδο με τις ΗΠΑ θα βρισκόμασταν εμείς σε ασθενή θέση. Νομίζω ότι θα πρέπει πραγματικά να δούμε αν μπορούμε να προωθήσουμε περισσότερο πολυμερές θέσεις και να αποφύγουμε τις δεμερείς σχέσεις με τις ΗΠΑ, οι οποίες τελικά δεν είναι αξιόπιστες. Έπειτα, πρέπει να δούμε ποια Ποιοι άλλοι εταίροι εξίσου σημαντικοί με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να συμμορφωθούν με τους κανόνες του ΠΟΕ. Οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν θέλουν να συμμορφωθούν με τον ΠΟΕ. Από την άλλη όμως η Κίνα θέλει να έχει το καθεστώς οικονομίας της αγοράς χωρίς να ακολουθεί τους κανόνες του ΠΟΕ. Ποιοι είναι λοιπόν οι αξιόπιστοι εταίροι αυτή τη στιγμή στο ύψος αν θέλετε των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι θα συμμορφώνονταν με τους κανόνες του ΠΟΕ. Και συμφωνώ με μια ερώτηση που ακούστηκε πριν από λίγο, πώς μπορούμε άραγε να μεταρρυθμίσουμε τον ΠΟΕ ώστε να λειτουργεί στην πράξη, να είναι αποτελεσματικός. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποιες παρατηρήσεις και ερωτήσεις σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Αρενά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται μια συγκεκριμένη στρατηγική θέλει να συσπυρώσει τις δυνάμεις της με την ομάδα φίλων του ΠΟΕ για παράδειγμα ή με άλλες δυνάμεις, με άλλους συμμάχους. Υπάρχει κάποια κοινή βάση προκειμένου να αναλάβουμε μια πρωτοβουλία. Και να αφορά τις εξελίξεις στις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς αξιολογείτε εσείς την κατάσταση. Τι χρόνο απαιτείται αυτή τη στιγμή όσον αφορά την όλη πρωτοβουλία των ΗΠΑ για τα αυτοκίνητα και τα εξαρτήματα αυτοκινήτων και όσον αφορά τη συζήτηση που γίνεται στην Γερουσία. Φαίνεται ότι υπάρχουν ορισμένοι που θέλουν να ανακτήσουν πλέον τις αρμοδιότητες αυτές, τις εμπορικές, έτσι ώστε να περάσουν τελικά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ στις βουλές, στην ομοθετική δύναμη, στην κοινοβουλευτική δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών. Ποια είναι η δική σας η άποψη σε σχέση με τις κινήσεις που έχουν ξεκινήσει αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο της Αμερικής. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολλές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις ακούστηκαν. Η πρώτη ερώτηση ε, σε ό,τι αφορά το μηχανισμό επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ ε, και το κατά πόσο μπορούμε να δημιουργήσουμε εδώ μια πολυμερή προσέγγιση. Να σας πω ότι προς το παρόν δεν θεωρώ ότι υπάρχει τέτοια βούληση από την πλευρά του ΠΟΕ για κάτι τέτοιο. Νομίζω πως η σωστή προσέγγιση θα ήταν να δούμε το τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να βελτιώσουμε τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών, ειδικότερα τα του δευτεροβάθμιου διοικητικού οργάνου. Ε, και δεν μπορούμε εδώ βέβαια να κάνουμε χρήση του όρου δικαστές. Ε, μιλάμε απλά για μέλη του δευτεροβάθμιου διοικητικού οργάνου, γιατί εκεί βέβαια συμμετέχουν και μέλη από την πλευρά των ε, ΗΠΑ. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε εδώ με ένα δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο και τίποτα παραπάνω. η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λοιπόν διατεθειμένη να εξετάσει τρόπους με τους οποίους μπορεί να βελτιωθεί αυτός ο μηχανισμός και να συζητήσει από κοινού και με άλλους τέτοιες δυνητικές βελτιώσεις. Η Αμερικανική πάντως πλευρά δεν έχει επιδείξει ε, κάποια βούληση από την πλευρά της ε, προκειμένου να διαπραγματευτούμε αυτό το ζήτημα. Ο κύριος στόχος πάντως από τη δική μας πλευρά θα πρέπει να είναι να διατηρηθεί αυτή η διαδικασία δύο φάσεων στο επίπεδο του μηχανισμού επίλυσης διαφορών. γιατί ε, αυτό που ακούμε είναι ότι ένας από τους στόχους ε, των Αμερικανών είναι να αφαιρεθεί, να εξαλειφθεί η δεύτερη φάση της διαδικασίας του μηχανισμού επίλυσης διαφορών, δηλαδή του δευτεροβάθμου οργάνου, έτσι ώστε να υπάρχει μόνο μία φάση επίλυσης διαφορών, δεσμευτική. Πράγμα το οποίο ήταν ε, πάρα πολύ ε, βέβαια ε, ε, το οποίο έγινε ως ε, πρόταση την τελευταία στιγμή ε, και βασίζεται στο αμερικανικό μοντέλο ενώ ταυτόχρονα υπάρχει και αυτό το μοντέλο της ΕΓΚΑΤ όπου ακριβώς υπήρχε αυτή, αυτή μία φάση στο μηχανισμό επίλυσης διαφορών ε, χωρίς να έχει δεσμευτικά αποτελέσματα. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε μεν τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών χωρίς ωστόσο να θέσουμε ένα αμφιβόλο ε, τις βασικές αρχές όπως για παράδειγμα αυτό της ανεξαρτησίας ε, και θα κατά τις επόμενες εβδομάδες εμείς ε, θα αναλάβουμε κάποιες πρωτοβουλίες με εταίρους που έχουν την ίδια άποψη έτσι ώστε να επιτύχουμε κάποια πρόοδο σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Τώρα σε ό,τι αφορά το rulebook θα επανέλθω σε αυτό αργότερα. Τώρα σε ό,τι αφορά την Κίνα δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον στο επίπεδο του ΠΟΕ να ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση ό,τι αφορά το μηχανισμό επίλυση διαφορών χωρί τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε θα πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά το, την ερώτηση του κ. Σαλαφράνου και της κ. και σε ό,τι αφορά τις ελιές. Ε, πράγματι μας ανησυχεί πάρα πολύ αυτό το ζήτημα και θα πρέπει να εξετάσουμε λίγο τι τις ε, λεπτομέρειες αυτής της απόφασης όταν αυτή θα εκδοθεί γιατί βέβαια ε, δεν νομίζουμε ότι θα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά όπως αυτή ε, της υπόθεσης Μπομπάρντιο. Οπότε ε, θα δούμε ε, ακριβώς με ποιον τρόπο ε, θα επιβληθούν αυτοί οι δεσμοί έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να προσφύγουμε σε επίπεδο που εναντίον τους ε, θεωρώντας ότι πρόκειται για αντι ε, dumping Αλλά βέβαια εδώ θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε και το σύστημα CEP το οποίο είναι ευρύτερο και δεν καλύπτει δηλαδή μόνο ελιές. Ε, δεν θα θέλαμε σε κάθε περίπτωση ο ΠΟΕ βέβαια με αυτόν τον τρόπο να αρχίσει να εξετάζει ε, σιωπηρά αν θέλετε ή με αυτόν τον τρόπο επειδή ξεκινούμε τη συζήτηση για τις ελιές ε, ε άλλες ε, ενισχύσεις που εμείς δίνουμε και εντάσσονται μέσα στο Green Box. θεωρούμε πάντως πως υπάρχουν ευρύτατες συνέπειες και υπάρχει κατάχρηση από την πλευρά των Ηνωμένων ε, Πολιτειών ε, σε ό,τι αφορά την χρήση αυτών των ε, κανόνων, ότι δηλαδή εφαρμόζουν υψηλότερους δασμούς επειδή θεωρούν ότι πρόκειται για αντιτάμπικ. Οπότε αυτή, αυτή η επιβολή τέτοιων περιορισμών από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί μέρος του προβλήματος, αποτελεί μέρος του και όχι λύση. Τώρα, και η Γενική Διεύθυνση Άγκρη, ε, Επίτροπος Χόγκαν και Επίτροπος Μάλστον ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα και αυτό καταδεικνύει ότι και στο μέλλον σε ό,τι αφορά την, ε, την απαγόρευση των ενισχύσεων κυρίως στον στόχαστο βρίσκονται ε, οι, τα μετρα αντιντάμπινγκ και στο επίπεδο λοιπόν του CMP θα πρέπει να αποφύγουμε ε, την επιβολή κλαδικών και μόνο περιορισμών σε ό,τι αφορά τις ενισχύσεις, μόνο για παράδειγμα στον τομέα της γεωργίας. Γιατί θα ήταν δυνατόν να πολλαπλασιαστούν τέτοιου είδου ε, ενισχύσεις ε, κλαδικές. Για παράδειγμα υπάρχει μια χώρα η οποία θα μπορούσε, έχει, ήδη εφαρμόζει 40 κλαδικές τέτοιες ενισχύσεις σε επίπεδο Blue Box και βέβαια τέτοιου είδους ενισχύσεις μπορούν να αμφισβητηθούν από άλλους εταίρους. και κατά συνέπεια θα μπορούσαν να αποτελέσουν τέτοιου είδους ενισχύσει εύκολο στόχο για την εφαρμογή μέτρων αντιντάμινγκ. Οπότε θα πρέπει ε, να δούμε στην ε, νέα ε, πώς μπορούμε να περιλάβουμε περισσότερες ενισχύσει στο green, green box, ε, για παράδειγμα μέσω ενό οριζόντιου συστήματο. Καθώ το Άμπερ θα ήταν πολύ δυσκολότερο να, δηλαδή μια ευρεία προσέγγιση σε ό,τι αφορά ενισχύσει του τύπου Green Box θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να ε, βρεθεί στο στόχαστρο ε, μέτρων anti-dumping από την πλευρά Τώρα, περνάω στο ζήτημα της Ρωσίας η Ρωσία παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα. Και δεν βλέπουμε να υπάρχει διάθεση από τη ρωσική πλευρά να βελτιωθούν τα πράγματα. Υπάρχουν πολλές υποθέσεις που έχουν κινηθεί κατά της Ρωσίας στον ΠΟΕ πρόσφατα ε, και είναι για πρώτη φορά συμβαίνει το ένα νέο μέλος να βρίσκεστε στο στόχαστο τόσων υποθέσεων, δηλαδή να, κατηγορείτε για τόσα ζητήματα. Και παρότι έχασε παταγωδός πρόσφατα σε μια υπόθεση έσπια σε ό,τι αφορά το χοιρινό κρέα, αυτό που έκανε η Ρωσία αντιδρώντας ε, ήταν να ε, επιβάλλει Οπότε, εάν δεν υπάρξει λύση σε σχέση με αυτό το ζήτημα και η ρωσική πλευρά δεν κάνει αυτά που χρειάζεται ε, ούτως ώστε να συμμορφωθεί δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα εμείς με το να κινηθούμε εναντίον και των ε, νέων μέτρων που έχει επιβάλλει. Πάντως σε σχέση με τη Ρωσία είναι σαφές ότι θα μπορούσαμε να επιτύχουμε μια βελτίωση του εμπορίου μας με τη Ρωσία αλλά δεν βλέπουμε ε, κάποια θετικά ε, βήματα από δική του πλευρά. Και βέβαια από γεωπολιτική άποψη, λαμβάνοντα υπόψη τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία και πάλι δεν βλέπουμε καμία βελτίωση με τη Ρωσία. Τώρα, τα όσα είπε ο κ. Σάκη ό,τι αφορά την ανάγκη του να παραμείνουμε ενωμένοι, ναι, είναι σαφέ. Και σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, η οποία αναφέρθηκε από άλλους ομιλητές, και ε, το, τον κίνδυνο κλιμάκωση ε, της ε, διαμάχης εδώ μεταξύ ΗΠΑ και Κίνα, να πω καταρχήν ότι η Κίνα προσχώρησε στον ΠΟΕ το 2001 και τότε οι περισσότεροι εταίροι ε, ανησυχούσαν με την πρόσβαση που είχε πλέον η Κίνα στις ε, αγορές ε, και τότε είχε ζητηθεί από όλους τους εταίρους να υπάρξει εφαρμογή αυτού του ενιαίου εγχειριδίου κανόνα του rule book αλλά σήμερα είναι σαφές ότι το rule book αυτό δεν επαρκεί για να καλύψουμε τα θέματα με την Κίνα σε ό,τι αφορά την ενίσχυση, σε ό,τι αφορά τη μεταβίβαση της ε, ε, τεχνογνωσίας, ε, σε ό,τι αφορά τις κοινές επενδυτικές κοινοπραξίες και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν αυτό θα, πρέπει να αποτελέσει ένας από τους στόχους μας στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του ΠΟΕ. Και είναι κρίμα το ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, εφαρμόζουν κάποια μέτρα αυτή τη στιγμή τα οποία θεωρητικά προσπαθούν να τις προστατεύσουν από την Κίνα αλλά ουσιαστικά ε, μας αποδυναμώνουν όλους ε, συλλογικά εναντί της Κίνας. Αντί δηλαδή να αξιοποιήσουμε την τρέχουσα κρίση έτσι ώστε να πάμε στην καρδιά του κινέζικου συστήματος και να ζητήσουμε να αξιώσουμε μια μεταρρύθμιση από την Κίνα, με ε, την, ε, αυτήν την μεταστροφή που κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε και ουσιαστικά στρέφονται κατά των ιδιωτέρων τους, ε, αυτό υπονομεύουν τις προσπάθειές μας. Και σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της ΗΠΑ και Κίνας, ε, δεν ξέρω, ο πρόεδρο Τραμπ λέει ότι οι εμπορικοί πόλεμοι είναι εύκολοι, εύκολο να νικηθούν, αλλά νομίζω πω ο συγκεκριμένο εμπορικό πόλεμο θα είναι πολύ κακό για όλου. Ε, και δεν νομίζω ότι η Κίνα θα χάσει αυτό τον εμπορικό πόλεμο. Δεν θα είναι η Κίνα ο ηθημένο από του δύο. Οπότε εδώ ε, αδυνατό να αντιληφθώ τον στόχο εδώ των ΗΠΑ. Τώρα, είναι δύσκολο να αναλύσουμε τις άμεσες συνέπειες σε ό,τι αφορά τα προϊόντα τα οποία έχουν μπει και στο άμεσο στόχο από την δική μας ε, πλευρά. Αλλά τα αναλύουμε αυτή την περίοδο. Σε κάθε περίπτωση όμως, ε, σε ό,τι αφορά την, το παγκό, την παγκόσμια ατμόσφαιρα, αν θέλετε το παγκόσμιο κλίμα, γιατί υπάρχει και, υπάρχουν και θετικές και αρνητικές ε, προσδοκίε σε επίπεδο ακριβώ του παγκοσμίου εμπορίου, μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά δεν είναι θετικέ οι προσδοκίε. Ε, τώρα σε ό,τι αφορά το σχόλιο του Κρίστοφ Χέλνερ, σε ό,τι αφορά τις σκέψεις που θα πρέπει να κάνουμε σε σχέση με τις δράσεις που θα πρέπει να αναλάβουμε τώρα άμεσα τα επόμενα βήματα. Ε, εμείς δεν πρόκειται να προβούμε σε αντίπεινα, δεν χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο. Ε, προβαίνουμε σε αντίμετρα, αναλογικά, τα οποία βασίζονται στην συμφωνία των Εσέβιων, των εγγυήσεων, Γιατί αυτό κάνει ουσιαστικά με συγκεκριμένο τρόπο η Αμερικανική πλευρά και εμείς απαντούμε με τον ίδιο τρόπο. Και καλύπτουμε μόνο το 40% των μέτρων τα οποία έχουν επίπτωση σε εμάς. Και από εκεί και μετά. Ω προ το ποιε θα μπορούσαν να είναι οι δυνητικέ ε, συνέπειε αν χάσουμε μια τέτοια υπόθεση στον ΠΟΕΑ ή αν κερδίσουμε. Καταρχήν να πω ότι θα πρέπει να βρούμε μια λύση σε ό,τι αφορά το δευτεροβάθμιο ε, δικαιοδοτικό όργανο. Γιατί α, χωρίς αυτό δεν θα υπάρξει μια σχετική απόφαση. Ε, και βέβαια μια τέτοια απόφαση ούτως ή άλλως θα χρειαστεί αρκετό χρόνο. Αν χάσουμε πάντως θα είναι καταστροφικό κάτι τέτοιο, γιατί θα σημάνει ότι τα πάντα θα επιτρέπονται πλέον. Και από πλευρά χρονική συγκυρία ε, να πω πως η οριστική απόφαση σε επίπεδο ΠΟΕ θα εκδόταν ε, σε τρία χρόνια. Το συντομότερο. Ε, δηλαδή μετά από την, ε, με την, τρέχουσα θητεία του Πρόεδρου Τραμπ. Γιατί βέβαια δεν γνωρίζω αν θα ανανεώσει τη θητεία του ή όχι. Όσον αφορά τα ζητήματα πιο συστημικής φύσης, πέθεσε ο κύριος Σόλτς. Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Πρώτον, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ ότι το πιο ουσιαστικό διαρθρωτικό πρόβλημα είναι η Κίνα και οι φυστάμενες πρακτικές της Κίνας, οι οποίες δεν οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά τις ε, επιδοτήσεις και όσον αφορά τη μεταφορά τεχνολογίας και γι' αυτό το λόγο έχουμε στραφεί εναντίον της Κίνας για το ζήτημα αυτό. Παρότι υπάρχει μια πολύ δύσκολη κατάσταση με τη ΣΥΠΑ, έχουμε κρατήσει την τριμερή αυτή συνεργασία με τις Ηνωμένε πολιτείες και με την Ιαπωνία για τα ζητήματα τα οποία αναφέρατε. Και ξέρετε ότι έγινε και μια δήλωση στον τύπο, μια κοινή δήλωση τύπου, όπου ο πρέσβης Λαϊτάιζερ και η Επίτροπος Μάλστρομ, καθώς επίσης και άλλοι αξιωματούχοι που ήταν στο Παρίσι στις 31 Μαΐου, είπανε ότι θα πρέπει από κοινού να συνεργαστούμε προκειμένου να βελτιώσουμε το rule book, των αγχειρίδιων κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Όσον αφορά το ζήτημα των επιδοτήσεων καταρχάς, εκεί τα πράγματα δεν είναι επαρκή και σαφή σε αυτό το εγχείρητο κανόνων και δεύτερον ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με τη μεταφορά τεχνολογίας και με τα πνευματικά δικαιώματα και τρίτον ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα ζητήματα καθεστώτος οικονομίας της αγοράς και ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα το εφιστάμενο σύστημα του ΠΟΕ όσον αφορά τη διαφάνεια και όσον αφορά την κοινοποίηση. Γιατί και ως προς αυτό υπάρχουν πολλά μέλη τα οποία δεν τηρούν τους κανόνες περί κοινοποίησης. Πολλά πράγματα λοιπόν βλέπετε ότι ήδη κάνουμε. Κρατούμε ανοιχτή αυτή την άγουσα αν θέλετε. Και νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πλήρως όλο τα διαθέσιμα μέσα τα οποία έχουμε. Πάντως, αυτή τη στιγμή η υπουργική διάσκεψη όσον αφορά τις χώρες παραγωγής χάλιβα που θα λάμβανε χώρα στο Παρίσι υπό Προεδρία της Αργεντινής θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα το Σεπτέμβριο. Γιατί ουσιαστικά εδώ πέρα θέλουμε να έχουμε πλήρη δέσμευση όλων των συμμετεχόντων χωρών. Η Κίνα, για παράδειγμα, παρά τα μέτρα αυτά τα οποία ανακοίνωσαν οι Πολιτείες, προσπαθεί μέσω των μέτρων 2-3-2 να πετύχει την άρση των μέτρων αυτών ουσιαστικά. Νομίζω ότι τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποίησαμε εμείς στο παρελθόν δεν ήταν τα πλέον αξιόπιστα. Γιατί εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε επηρεαστεί πάρα πολύ περισσότερο από τους δασμούς των ΗΠΑ από ότι η Κίνα μέσω των μέτρων της κατηγορίας 2 Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου την κατάσταση αυτή και ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσει η Κίνα σε σχέση με την υπερπαραγωγή χάλιβα. Τώρα, ...δε αυτή που ακούστηκε ότι η κρίση αυτή η εμπορική θα μπορούσε να αποτελέσει και ευκαιρία. Δεν διαφωνώ. Στα πλαίσια κρίσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποιο είναι το πρόβλημα και ποιοι είναι οι στόχοι των εμπλεκόμενων εταίρων εφόσον το γνωρίζουμε αυτό, μπορούμε και να διέλθουμε από την κρίση σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι πριν. Εν προκειμένου όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρουμε να καταλάβουμε πρώτον. Εγώ από προσωπικής πλευράς για παράδειγμα δεν είμαι σίγουρος τελικά για το ποιε είναι, ποιοι είναι οι πραγματικοί στόχοι του Προέδρου Τραμπ. Έχει άραγε σαφείς στόχους μέσα από την πολιτική του. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι πρώτον να προωθήσουμε ένα νέο TTIP ή να αναστήσουμε, αν θέλετε, τις προηγούμενες διαπραγματεύσεις TTIP. αυτό δεν θα οδηγήσει πουθενά. Για ποιο λόγο άραγε μπλοκαρίστηκαν οι προηγούμενες διαπραγματεύσει TTIP. Ξέρετε ότι με την προηγούμενη Αμερικανική κυβέρνηση, όπου λογικά θα είχαμε καταλήξει σε μία λύση όσον αφορά τη συμφωνία αυτή και τις σχετικές διαπραγματεύσει τελικά δεν τα καταφέραμε, είναι αδύνατο ποτέ να τα καταφέρουμε με αυτή την ε, κυβέρνηση. Και ας μην ξεχνάμε ότι 15 συναντήσεις ε, ή α, τηλεφωνικές κλήσεις, αν θέλετε, ή τηλεδιασκέψεις μάλλον, γίνανε μεταξύ της Επιτρόπου Μάλστρομ και του Υπουργού Εμπορίου ΡΟΣ των Ηνωμένων Πολιτειών και εμεί σε κάθε περίπτωση, σε κάθε μία από τις επαφές αυτές, Ήμασταν έτοιμοι να προτείνουμε πιο ευνοϊκά δασμολογικά μέτρα σε σχέση με τις ΗΠΑ αν μας, αν μας βγάζανε από τον κατάλογο δασμολογικών ε, ε, μαλλοτελουνιακών δασμών που έχουν επιβάλει. Σίγουρα στη Γεωργία θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να κάνουμε παραχωρήσεις. Πάντως ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε παραχωρήσεις σε πάρα πολλά προϊόντα. Ήταν άκαμπτοι, άκαμπτοι από την Αμερικανική πλευρά. Ο Υπουργός Εμπορίου Ρώσ των ΗΠΑ μας πίεζε κάθε φορά να αποδεχθούμε πολύ σκληρούς δασμούς στο χάλιβα και στο αλουμίνιο με μείωση τελικά των εξαγωγών μας και μας έλεγε ότι αυτό θα έπρεπε να το καταπιούμε πολύ απλά. Και ότι υποτίθεται ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα βρισκόταν μία λύση και ότι θα υπήρχε και μία εξηλαίωση από τη δική μας την πλευρά γιατί υποτίθεται ότι έχουμε αμαρτήσει στα μάτια των ΗΠΑ. Πάντως νομίζω ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τρόποι εξέβρεσης λύσης. Αυτός μην το ξεχνάμε για οποιοδήποτε πρόβλημα, για οποιοδήποτε προϊόν, ακόμα και για τα αυτοκίνητα. Αλλά δεν μπορούμε προφανώς εμείς προκειμένου να βρούμε λύση, να κάνουμε μονομερείς μόνο εκχωρήσεις και παραχωρήσεις. Και η προσέγγιση εκείνη η οποία έχει να κάνει με την νεοθέτηση παράνομων εμπορικών κανόνων και που Ζητάει εν συνεχεία ως τακτική να καταβληθούν λίτρα προκειμένου να αποσυρθούν οι παράνομοι αυτοί κανόνες, ε, αυτό δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε σε καμία περίπτωση. Προφανώ δεν μπορούμε να δεχθούμε τέτοιου εκβιασμούς. Εμείς θέλουμε να μπορούμε να συμμετέχουμε σε λογικές ε, συζητήσεις, σε ένα πνεύμα θετική συνεργασία, αλλά όχι με δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι μα, χωρί απειλέ και χωρί. Ε, Τώρα, σε σχέση με τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις του κυρίου Σαλαφράγκα, όσον αφορά τις ποσοτικές επιπτώσεις όλων αυτών των μέτρων, κοιτάξτε, είναι σαφές ότι όλα αυτά τα μέτρα θα είναι επιζήμια και κυρίως για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για το Χάλιβα, για παράδειγμα, το λένε όλοι. Αυτό θα είναι κυρίως επιζήμια για τις Ηνωμένες Πολιτείες θα υπάρχουν κάποιες αν θέλετε επιφανειακές βελτιώσεις σε επίπεδο Αμερικής όσον αφορά την παραγωγή χάλιβα, αλλά σε βάθος χρόνου θα καταργηθούν πάρα πολλές θέσεις απασχόλησης. Και δεν νομίζω ότι θα μπορούσε ποτέ μέσω των μέτρων αυτών ο κύριος Τραμπ να αποκαταστήσει την πολύ ψηλή ανεργία η οποία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80 σε πολιτείες όπως η Αριζόνα κτλ. Δεν είναι τέτοια μέτρα αυτά τα οποία θα βοηθήσουν την κατάσταση των ΗΠΑ. Ξέρετε ότι στο παρελθόν και σε τέτοιες περιπτώσεις χρησιμοποιώντας τις ρήτρες διασφάλισης έχουμε καταφέρει να νικήσουμε πολλές υποθέσεις ε, στον ΠΟΕ και σίγουρα όχι μόνο για το χάλιβα αλλά και για τα αυτοκίνητα και τα εξαρτήματά τους τα μέτρα τα οποία λαμβάνουν οι μονές πολιτείες ήταν επιζήμια για τη, δικά τους, για τη δική τους την οικονομία. Τώρα για την ναύτα και πιο συγκεκριμένα πάλι για προϊόντα όπως τα αυτοκίνητα και τα εξαρτήματα αυτοκινήτων, ξέρετε ότι η ενσωμάτωση των προϊόντων αυτών αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στην οικοδόμηση της ναύτα. Και αυτόν γέννη ήταν θετικό για όλους. Ε, είναι σαφές ότι έχουν έλλειμμα εμπορικό οι Ηνωμένες Πολιτείες, και σαφώς υπάρχουν πολύ ολοκληρωμένες αλυσίδες αξίας στα πλαίσια της ναύτα και δεν μπορούμε ποτέ να πούμε ότι η επίδραση της ναύτα ήταν αρνητική σε παγκόσμιο επίπεδο. Και όσον αφορά το Μεξικό και τον Καναδά, πάλι εκεί πέρα θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση από εκείνη την πλευρά, αλλά μην ξεχνάμε ότι Ενδεχομένως να πρέπει να υπάρχει εδώ πέρα μία ρήτρα αναστολή sunset clause για μία επαναδιαπραγμάτευση κάθε πέντε χρόνια της συμφωνίας αυτή, Αλλά ούτε το Μεξικό, το Καναδάς, ούτε άλλοι θέλανε ποτέ να ισχύσει τελικά κάτι τέτοιο και ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελε μια τέτοια περιοδική τακτική αναθεώρηση της ναύτα. Πάντως το ζήτημα των αυτοκινήτων και των εξαρτημάτων τους που θέσατε σαφώς έχει να κάνει και με την ναύτα και το καλό είναι ότι για τα προϊόντα τουλάχιστον αυτά έχουμε καλή συνεργασία με το Μεξικό και τον Καναδά. Τώρα, όσον αφορά τα αντίπεινα, ένα άλλο σχόλιο το οποίο ακούστηκε, δεν έχουμε υιοθετήσει ούτε πρόκειται να υιοθετήσουμε αυτή τη στιγμή προωθούμε μέτρα αντισταθμιστικά, μέτρα εξισορροπητικά. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε κάπως την ψυχοσύνθεση του κύριου Τράμπα. Σε καμία περίπτωση πάντως δεν θα πρέπει να ρίξουμε περισσότερο λάδι στη φωτιά αυτή τη στιγμή. Και δεν θα πρέπει εμείς απέναντι σε μια τέτοια στάση βέβαια να φανούμε αδύναμοι. Αν δεν αντιδράσουμε καθόλου, τότε το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχουμε μια αέναη διαδικασία επιβολής νέων μέτρων και νέων κυρώσεων από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να περασπίσουμε πάση θυσία τα συμφέροντά μας και προφανώς μέτρα τέτοιου είδους δεν είναι θετικά σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά θα πρέπει εμείς να καταφέρουμε να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τη σέβονται και ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να αντιδράσει. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημα της κυρίας Αρενά, το ερώτημα της κυρίας Αρενά που έχει να κάνει με τις διμερείς σχέσεις. Μα οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ήδη αντιδράσει. Το TTIP αυτή τη στιγμή δεν απασχολεί καθόλου τις Ηνωμένε Πολιτείε, ούτε τίθεται εκ νέου ως πρωτοβουλία που θα μπορούσε να επαναπροωθηθεί. Αν γίνουν κάποια θετικά διαβήματα από τις Ηνωμένε Πολιτείε, εμείς θα τα αποκριθούμε. Αλλά περιμένουμε ακόμα να δούμε ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση, μονομερής, διμερής ή πολυμερής. Προσωπικά νομίζω ότι ε, θα ήταν το καλύτερο να συνεργαστούμε με άλλες μεγάλες δυνάμεις οι οποίες σκέφτονται και λειτουργούν όπως εμείς. Τώρα, όσον αφορά άλλε χώρε, συνεργαζόμαστε πολύ καλά με την Ιαπωνία, τον Καναδά, το Μεξικό, την Κορέα. Ε, έχουμε συμφέρον λοιπόν να προωθήσουμε αυτές τις σχέσεις. Και να απαντήσω και στην τελευταία ερώτηση του Προέδρου του κ. Λάγκε Μας ρωτήσατε για την ημερομηνία επιβολής των μέτρων αυτών. Κοιτάξτε, το σχέδιο του κυρίου Τραμπ είναι σαφέστατο κάτι να απόψή Αυτό το οποίο προσπαθεί να πετύχει αυτή τη στιγμή είναι για εσωτερικούς εκλογικούς λόγους να καταφέρει να εγκρίνει τα μέτρα αυτά για τα αυτοκίνητα και τα εξαρτήματα αυτοκινήτων πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Αυτό το χρονοδιάγραμμα πιστεύω λοιπόν ότι θα ακολουθήσει. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει και εμείς ε, γρήγορα να αντιδράσουμε. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο αυτή τη στιγμή για να εστιαστούμε πολύ συγκεκριμένα στο ζήτημα των αυτοκινήτων. Θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να λύσουμε αυτό. Πάντω το ζήτημα είναι, παρουσιάζει αρκετές πολυπλοκότητες. Ενδεχομένω να μην γνωρίζετε ότι η ευρωπαϊκή αυτοβιομηχανία και η παραγωγή της στις ΗΠΑ εξάγει ως τον ίδιο αριθμό αυτοκινήτων που εξάγει προς την Κίνα για παράδειγμα με αυτόν τον αριθμό που εξάγει στι ΗΠΑ. Η παραγωγή τους λοιπόν και οι εξαγωγέ του προ τι ΗΠΑ είναι εξίσου σημαντική με αυτή προς τον υπόλοιπο κόσμο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το ζήτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να εξεταστεί και από πολιτική ε, πλευρά και θα πρέπει και με τους επιχειρηματίες αλλά και με, τους, και με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να αποτιμήσουμε τον κίνδυνο των μέτρων αυτών και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποφύγουμε εμείς με τη δική μας τη στάση να οδηγηθούμε σε αρνητικά αποτελέσματα. Νομίζω ότι μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα πρέπει να δούμε πώς τα μέτρα αυτά για τα αυτοκίνητα μπορεί να επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις μας με την Κίνα Επί του παρόντος πάντως σίγουρα η στάση μας, η εμπορική επέναντι στην Κίνα για τα αυτοκίνητα δυσχεραίνεται εξαιτία της στάσης των ΗΠΑ. Προσπάθησα να απαντήσω στις περισσότερες τουλάχιστον ερωτήσεις. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα παραπάνω. Είναι σαφές πάντως για μένα ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και πολύ αποφασιστικοί. Το χειρότερο, αν θέλετε, σενάριο θα είναι να καταφέρουμε εμείς να διασπαστούμε τα κράτη-μέλη δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να διχαστούμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Ζανλίκ. Και ελπίζω να μην είναι τελευταία φορά που θα έχουμε μαζί σου αυτή τη συζήτηση για την κατάσταση και την αντίδρασή μας. Έχεις δίκιο ότι το σημαντικότερο είναι να είμαστε ενωμένοι ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα η απάντηση στο America First είναι Ευρώπη Ενωμένη. Okay. So, the uh, next item... Το επόμενο σημείο So, Straight away. So, Αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη έχει σχέση με το προηγούμενο τη εμπορική σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση είπα. Έχει να κάνει με την προστασία της βιομηχανία μας από την εξοεδαφική εφαρμογή ορισμένων νόμων που έχουν θεσπιστεί από μια τρίτη χώρα. Σε ισχύ Έχουμε μία ε, νομοθεσία ήδη από το 1996. Το 2005, νομίζω, έγινε μια απόπειρα αναδιατύπωσης ε, της ε, νομοθεσίας αυτής. Α, εντάξει. Αργότερα ήτανε. Τους έγινε μια απόπειρα αναδιατύπωση της ε, πολύ παλιά αυτή νομοθεσίας, την οποία για να σας ε, το πω αυτό εν μόνο μια χώρα και μόνο μία περίσταση αναφερόταν, η Κούβα. Και εξοεδαφική εφαρμογή νόμων. Συγκεκριμένα κυρώσει και πρόστιμα. Εμπάργκο πάνω στην Κούβα. Έχει αλλάξει όμως η κατάσταση άρδιν έκτοτε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε με κατεξουσιοδότηση πράξη για τροποποίηση αυτής της παλιάς νομοθεσίας σε ό,τι αφορά την εξοδοφική εφαρμογή των ενδεχόμενων κυρώσεων και της επίπτωσης αυτών. Συγκεκριμένα για τις ε, κυρώσεις ε, και για τον αντίκτυπο που είχε αποχώρηση τον ΙΠΑ από τη συμφωνία με το Ιράν. Επίσης, ξανά στο τραπέζι και το θέμα της αναδιατύπωσης. Είναι όμως πολλά τα πράγματα. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς για ποιο λόγο. Ελπίζω να έχουμε κάποιες διευκρινήσεις σήμερα για να ξανακατέβει από τα σύννεφα και να μπει στο τραπέζι αυτή η αναδιατύπωση. Αυτά ως μια σύντομη εισαγωγή. Θα ακούσουμε τον εισηγητή μας, τον David Μάρτιν τώρα. Θα μας τα πει καλύτερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά και έχετε δίκιο ότι σχετίζεται στενά με το προηγούμενο θέμα αυτό και έχει να κάνει με τη μονομερή προσέγγιση των ΗΠΑ. για τις πράγματα για την αναδιατύπωση αυτού του κανονισμού ε, που είναι από τη δεκαετία του 1990 από το 1996 και ποτέ ουσιαστικά δεν έχει χρησιμοποιηθεί όμως ε, χρησιμοποιήθηκε αποτρεπτικά ε, και δεν επέβαλε η, ε, η δεν επέβαλαν οι ΙΠΑ τις κυρώσεις που θα είχαν επιβάλει σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κούβα. Επομένως είχε κάποια αποτρεπτική ισχύ και όπως είπατε πράγματι υπήρξε επίσημη πρόταση αναδιατύπωσης της υπνότουσας αυτής νομοθεσίας ε, το 2015 συγκεκριμένα. Εγώ διατύπωσα το 2015 μία, μάλλον ε, κατέθεσα ένα σχέδιο έκθεσης, αλλά δεν προχώρησε διότι η νομική υπηρεσία, συγκεκριμένα οι νομικές υπηρεσίες των τρίτων, ε, των τριών θεσμικών οργάνων δεν συμφώνησαν σε ό,τι αφορά την τεχνική της αναδιατύπωσης και κόλλησε το θέμα στο Συμβούλιο. Και εσείς, Μπέρντ και εγώ είχαμε γράψει στην Μογκερίνη το Φεβρουάριο, θυμάστε καλά, και είχαμε ζητήσει η ΕΕΔ ε, να μας πει κατά πόσον θα θέσει υπόψη της Κομισιόν ένα αίτημα για κατάθεση μιας πρότασης. Είπε η κυρία Μαγκερίνη ότι ξέταζε διάφορες επιλογές. Δεν μας οδήγησε αυτό βέβαια όπως καταλαβαίνετε προς τα εμπρός. Τώρα, ε, για το τι συμβαίνει τώρα. Όπως είπατε, ο πρόεδρος Τραμπ τον προηγούμενο μήνα ανακοίνωσε ε, την αποχώρηση της ε, χώρας του από το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράση με το Ιράν και οι αρχηγοί κρατών και μέσα της Ευρωπαϊκής αποφάσισαν να επανεργοποιήσουν το καθεστώς που θα τους επιτρέπει να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους σε σχέση με το Ιράν και είμαστε στην κατευθότηση πράξη. Προτείνεται να περιληφθεί αναφορά σε αυτή την, ε, σε αυτή την νομοθεσία των 96 για τις κυρώσεις ε, των ΙΠΑ. Will the Commission present a new proposal? Έχουμε λοιπόν αυτό εδώ το block and start. Θα πρέπει να δούμε όμως ε, ποια νομική μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί και τώρα έρχομαι στην ουσία Υπάρχουν εταιρείε που δραστηριοποιούνται ε, με, στο Ιράν, τραπεζικές συναλλαγές, προϊόντα πετρελαιοειδή, μεταφορές, ε, ε, οχήματα δικού σκοπού κτλ. Δεν ξέρω αν οι ε, Κομισιόν και οι ΕΕΔ έχουν αξιολογήσει τι αντίκτυπο θα είχε απόφαση του Τραμπ για τις επιχειρήσεις μας. Με βάση τις ε, πληροφορίες που έχω, ίσως η ΕΕΔ όμως έχει πιο επικαιροποιημένε πληροφορίες, μιλάμε για 16 Βρετανικές, για, με 60 μάλλον Βρετανικές, 30 Γερμανικές, 35 Γερμανικές, 21 Ιταλικές, εταιρείε και ολιγάριθμες άλλες εταιρείε από άλλα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε καλό βαθμό ήδη θεωρεί ότι αυτό το blocking statute δεν θα μπορούσε ίσως παρά να έχει περιορισμένη ε, επίπτωση, ιδίω ό,τι αφορά το διεθνέ τραπεζικό σύστημα και την έκθεση μεγάλων συστημικών τραπεζών στο διεθνέ χρηματοπιστωτικό σύστημα και στι συναλλαγέ με δολάρια. Ε, και πάντα έχοντας υπόψη και την προηγούμενη συζήτηση, νομίζω πρέπει να έχουμε υπόψη ότι εδώ έχουμε μια διαφορετική αμερικανική κυβέρνηση από ό,τι είχαμε τότε, το 1996 δηλαδή. Και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την υλοποίηση, αν ε, δούμε ε, τις δράσεις προτείνεται να, προτείνεται να λάβει η Κομισιόν, δεν ξέρω αν θα έπρεπε να υπάρχει και ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο για την κάλυψη αποζημιώσεων, ε, για την αντιμετώπιση των ζημιών που θα προκύψουν. Και νομίζω ότι αυτό το blocking statute, ε, το κανόνας παρεμπόδισης, ε, θα μπορούσε να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο ώστε να μπορέσουν να βασιστούν σε αυτό οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις Εντάξει, μπορεί να είναι απλά ένα χαζαπλάστ σε μια μεγάλη πληγή, αλλά τέλος πάντων, έστω μια προσπάθεια να γίνει τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον κανόνα παρεμπόδιση στο μέλλον, θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματικός, θα μπορούσε να γίνει μια συζήτηση, όπως την πρώτη φορά με τα θεσμικό όργανα, που βέβαια δεν ήταν και τόσο ενθαρρυντική, αλλά δεδομένων των σημερινών περιστάσεων θα μπορούσε να είναι κάτι χρήσιμο η οι Υπουργοί Οικονομικών ε, ε, Γερμανίας, Αγγλίας, Γαλλίας ζήτησαν εξαίρεση από την εξοδαφική εφαρμογή. Μάλλον θα πάρουν αρνητική απάντηση, αλλά δεν ξέρω τι απάντηση υπήρχε και αν οι ευρωπαϊκέ εταιρείε εξαιρεθούν ή όχι είναι ένα θέμα που θα ήθελα να το συζητήσουμε και μια απάντηση να λάβω. Ευχαριστώ που σοβαρά τα ερωτήματά σα για την πρόταση και για την κατάσταση όσο έχει αυτή τη στιγμή. Έχουμε τρεις εμπειρογνώμονες τώρα που θα προσπαθήσουν να ε, ρίξουν λίγο φως στο σκοτάδι σε ό,τι αφορά την αναδιατύπωση. Και ίσως να δώσουν και κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματα για την ε, σημερινή κατάσταση. Θα δώσω καταρχάς το λόγο για 3 πεντε λεπτά. Θα αρκετός χρόνος νομίζω είναι. Στον David Gear που είναι επικεφαλής του τμήματος επιβολής κυρώσεων και προστήμων από την ΕΙΕΔ. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να σε ενημερώσουμε για το σημαντικό αυτό ζήτημα. Όπως υπόθηκε, θα ήθελα να σας δώσω κάποιες λεπτομέρειες για το γενικότερο πλαίσιο των εξελίξεων αυτών. Όπως ξέρετε, ο πρόεδρος Τραμπ στις 8 Μαΐου ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα αποχωρήσουν από το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης και παράλληλα δήλωσε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε θα επαναθεσπίσουν τις κυρώσεις αυτές οι οποίες είχαν καταργηθεί στα πλαίσια του νέου αυτού σχεδίου με το Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε αμέσω ενωμένη στάση, με τρόπο σαφέστατο, είπα ότι εκπρόσωπος προχώρησε σε δήλωση, περαιτέρω δηλώσεις γίνανε σε μια ειδική συνεδρίαση μεταξύ της είπα εκπροσώπου και των Υπουργών Εξωτερικών της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου και του Υπουργού Εξωτερικών Ζαρίφ του Ιράν. Και έπειτα στις 16 Μαΐου στη Σύνοδο της Σόφιας έγινε σαφής δήλωση ενότητας και αποφασιστικότητας από την ευρωπαϊκή πλευρά προκειμένου να διασωθεί το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης με το Ιράν το οποίο βέβαια παρουσιάζει ένα σημαντικό στρατηγικό ενδιαφέρον για μας και γενικότερα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τον υπόλοιπο κόσμο για την μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Παράλληλα, η άρση των κυρώσεων θεωρήθηκε από τους ηγέτες σαν απόσπαστο στοιχείο του σχεδίου αυτού και ανακοινώθηκε αυτό το λόγο ότι θα καταβάλουμε προσπάθειες προκειμένου να διατηρήσουμε τα ωφέλη της άρσης των κυρώσεων μαζί με τα άλλα μέλη της κοινής Επιτροπής και στο πλαίσιο όσων προβλέπονται από, την σχετική, από το σχετικό ψηφίσμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Όσον αφορά την επαναθέσπιση των κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών, ακόμα δεν γνωρίζουμε ακριβώς την εμβέλεια που θα έχουν. Πάντως, το όλο το ύφο το έθεσε ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος μίλησε για κυρώσεις πολύ μεγάλης εμβέλειας, πολύ γενικές κυρώσεις, μεγαλύτερες ενδεχομένως από ό,τι στο παρελθόν. Ο Υπουργός Εξωτερικών Πομπέιου επίσης το επανεβεβαίωσε αυτό στο λόγο του για τις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν και ο Υπουργό Εξωτερικών Μαντέλκα επίση αναφέρθηκε σε αυτό. Δύο περίοδοι εντοπίστηκαν, πρώτον από τις 6 Αυγούστου και η δεύτερη από τις 4 Νοεμβρίου και καλύπτουν οι χρονικές αυτές τις περίοδοι τα διαφορετικά είδη κυρώσεων που θα επαναεπιβληθούν από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Θα πρέπει να γνωρίσουμε ως προς αυτό ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε με τρεις εξαιρέσει ουδέποτε προχώρησαν σε άρση των πρωταρχικών βασικών τους κυρώσεων. Οπότε βασικά μιλάμε για την επανεγκαθίδρυση των δευτερογενών, θέλετε, κυρώσεων των κυρώσεων δεύτερης βαθμίδας. Και εδώ πέρα αναφερόμαστε σε ζητήματα που έχουν να κάνουν επίσης και με την πολιτική αεροπορία, με την κυκλοφορία των επιβατών και ούτω καθεξής. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, μετά τη συνεδρίαση της Σόφιας 18 Μαΐου ήταν να κοινώσει μια δέσμη μέτρων προκειμένου να εμφυσίσει νέα εμπιστοσύνη στο σχέδιο αυτό και έτσι ξεκίνησε εκ νέου η ε, παγκόσμια, συγγνώμη, η επίσημη διαδικασία προκειμένου να προχωρήσουμε περισσότερο με τον κανόνα παρεμπόδισης και προκειμένου να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε περισσότερα μέτρα οικονομικής εμπιστοσύνη με το Ιράν, καθώς επίσης και περισσότερα μέτρα οικονομικής δραστηριότητας σε συνεργασία με το Ιράν. Αυτά επίσης έγιναν παράλληλα με την έκκληση που έγινε προς τα κράτη-μέλη να ασχοληθούν περισσότερο με τραπεζικές μεταφορές προς την Κεντρική Τράπεζα των, του Ιράν. Μολονότι οι κυρώσεις αυτές δεν έχουν επιβληθεί εκ νέου, βλέπουμε ότι παρόλα αυτά έχουν αρχίσει να επηρεάζουν το εμπόριο και τις επενδύσεις με κάποιους βασικούς επενδυτές. Η Total, για παράδειγμα, που είναι βασικός επενδυτής στον ε, τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου ανακοίνωσε ότι θα φύγει από τη χώρα αυτή εκτός και αν βρεθεί μια εξαίρεση για αυτή. Και αν λάβουμε υπόψη την έκθεση των τραπεζών και του χρηματοπιστωτικού συστήματος στις ΗΠΑ και αυτός ο κλάδος ο χρηματοπιστωτικός θα ζημιωθεί πολύ σοβαρά. Δεν έχουμε συγκεκριμένε λεπτομέρειες, πάντως είχαμε έρθει σε επαφή και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με διάφορους επιχειρηματίες σε όλους τους κλάδους, προσπαθώντας να έχουμε μια πιο σφαιρική εικόνα του πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Θα πρέπει βέβαια να γνωρίζουμε ότι ο τραπεζικός και χρηματοπιστωτικός τομέας ήταν ήδη τομεί, κλάδοι, όπου υπήρχαν αρκετέ δυσκολίε, επειδή υπήρχε ήδη ο φόβο κυρώσεων από τι ΗΠΑ και κάποιε ανησυχίε όσον αφορά την διαφάνεια του ίδιου του Ιρανικού του χρηματοπιστωτικού συστήματο, πριν από τις τελευταίες αυτές εξελίξεις υπήρχαν όλες αυτές τις ανησυχίες. Πέρα από τις δηλώσεις λοιπόν που έκανε η ΥΠΑΤΗ εκπροσώπος, καθώς επίσης και τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεχίζουμε τις προσπάθειες προκειμένου να διατηρήσουμε τα ωφέλη από την άρση των κυρώσεων και μέσω τεχνικών συζητήσεων σε εσωτερικό επίπεδο αλλά και με το Ιράν και με άλλους όμως εταίρους προκειμένου να καταφέρουμε τελικά να αφήσουμε κάποιες προτάσεις σε βασικούς τομείς και σε ζητήματα όπως ο τραπεζικός τομέας ή το πετρέλαιο. Βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία και προφανώ ο κανόνα παρεμπόδιση αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο στι όλε τι συζητήσει που γίνονται για το εμπόριο και τι επενδύσει. Σα ευχαριστώ. Uh, η κυρία Μόνικα Έγξη, η ε, επικεφαλή τη μονάδα για την ε, Μέση Ανατολή, είναι επόμενη ομιλητρία μα. Ε, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και θα προσθέσω λίγα στα όσα είπε μόλις τώρα ο συνάδελφος ως προς την ανάγκη του να συνεχίσουμε τις επαφές μας σε ό,τι αφορά τα εμπορικά ζητήματα με το Ιράν και σκοπεύουμε να μεταβούμε εκεί την επόμενη εβδομάδα στο πλαίσιο ενό διαλόγου σε ό,τι αφορά εμπορικά και γεωργικά ζητήματα αλλά και ε, υγειονομικά και φυτο ε, θέματα αλλά και ζητήματα ε, διαλόγου και ένα διαλόγο σε ό,τι αφορά ζητήματα βιομηχανίας. Είχαμε συναντηθεί το 2016 σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων τον Νοέμβριο μάλιστα εκείνο το ετούσε μετά από 10 έτη ε, κανένα είδου επικοινωνία σε ό,τι αφορά ε, εμπορικά ζητήματα. Και εκεί είχαμε εντοπίσει μια σειρά από ζητήματα τα οποία ενδιαφέραν και το Ιράν και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, η ε, επανένταξη του Ιράν μέσα στην παγκόσμια αγορά. Εμεί είχαμε υποστηρίξει και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την προσχώρηση του Ιράν στον ε, ΠΟΕ, γνωρίζοντα βέβαια ωστόσο από το γεγονό ότι ε, μπλοκάρεται από το γεγονό ότι δεν είναι δυνατόν να διοριστεί ένα πρόεδρο αυτή τη ομάδα εργασία. Ε, Πάντω, εμεί θέλουμε να συμμετάσχει στο πολυμερέ εμπορικό σύστημα το Ιράν και έχουμε καταδείξει την πρόθεσή μα να το κάνει στην πράξη. Επίση, ε, θέλουμε να βελτιωθεί η διαφάνεια και να διευκολυνθεί το εμπόριο. Αλλά βέβαια το. Οι προσπάθειες που γίνονται είναι περιορισμένες γιατί βέβαια παραμένει μια κρατική οικονομία από εκεί και μετά υπάρχουν και ζητήματα βέβαια που αφορούν το ίδιο το εσωτερικό σύστημα ε, του Ιράν, για παράδειγμα το τραπεζικό του ε, σύστημα, όπου υπάρχει κάποια έλλειψη διαφάνεια και είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε μαζί του. Ε. Υπάρχει, ένας, υπάρχει σημαντική τεχνική αλλογή την οποία μπορούμε να παράσχουμε και θα έρθουμε σε επαφή με το Διεθνέ Εμπορικό Κέντρο έτσι ώστε να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τις προσπάθειές τους έτσι ώστε να βελτιωθούν για παράδειγμα τα ε, πρότυπα, τα τεχνικά ή τα πρότυπα SPS του Ιράν. Τέλος θα ήθελα να αναφέρω και τις επενδύσεις. Υπάρχουν μία σειρά από κράτη-μέλη τα οποία έχουν διμερείς συμβάσεις επενδύσεων με το Ιράν και νομίζω πως αυτό ήδη καταδεικνύει ότι οι δικές μας επιχειρήσεις ε, προστατεύονται ε, σε εκείνη την αγορά. Το Ιράν έχει δείξει κάποιο ενδιαφέρον ω προ τη σημασία Προστασία των Επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά μα. Και θα προβούμε σε αυτή τη συζήτηση, αλλά το ε, πιο σημαντικό βήμα σε εμπορικό επίπεδο είναι η προσχώρηση του Ιράν στον ε, ΠΟΕ. Ε, θα συνεχίσουμε λοιπόν τι επαφέ μα και, το... και τη δέσμευσή μα έτσι ώστε να καταδείξουμε ότι το γεγονό ότι οι ΗΠΑ προέβησαν σε μονομερή μέτρα δεν σημαίνει ότι εμείς δεν θέλουμε να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε ε, τα ωφέλη από την κατάργηση ε, των ε, κυρώσεων. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος, η κυρία Αλίνα Νάντερ από την Μονάδα για την Επιβολή Κυρώσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρώτα. Καλημέρα σε όλες και όλους και για μένα είναι χαρά που βρίσκομαι εδώ για να σας ενημερώσω για αυτά τα οποία ήδη ε, προανέφεραν οι συναφοί μου ως ένα από τα μέτρα τα οποία ενεργοποίησε η Κομισιόν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπίσει την απόφαση της ε, των ΗΠΑ για αποχώρηση από το κοινό ολοκληρωμένο για να με το Ιράν. Γνωρίζετε το ιστορικό, δεν θα ε, το επαναλάβω. Αυτό που θέλω όμω να σα υπενθυμίσω και αναφέρθηκε άλλωστε είναι ότι ο κανόνα παρεμπόδιση Broken ε, το 1996 μαζί με την πολιτική πίεση και την καταγγελία στο πλαίσιο που ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικό μέτρο ώστε ε, ΕΠΑ να μην εφαρμόζονται φθαρογενείς κυρώσεις ό,τι αφορά την Κούβα τότε σε ευρωπαϊκούς οικονομικούς φορείς. Και αυτό εξηγεί γιατί αυτός ο κανόνας ε, παρέμεινε σε πνότουσα κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Δεν χρειάστηκε να εφαρμοστεί, ε, χρησιμοποιήθηκε σε δυτικές διαφορές επίπεδο κρατών μελών, όμως δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλη κλίμακα γιατί δεν υπήρχαν υποθέσεις μεγάλης κλίμακας. Και αυτό θα ήταν καλό να το έχουμε υπόψη. Εν συντομία θα σας πω πώς ε, φτάσαμε στην πρόταση εξουσιοδότηση ε, πράξη που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι περιλαμβάνει το παράρτημα. Είπατε κι εσείς ότι ο κανόνας παρεμπόδισης από το 1996 αφορά την Κούβα, τις κυρώσεις δηλαδή τον είπα στην Κούβα. Μία πολύ σύντομη μια στο Ιράν έγινε με μία μόνο νομική πράξη. Τι έχουμε κάνει τώρα. Έχουμε εξετάσει όλες τις δευτερογενείς κυρώσεις των ΗΠΑ που ήρθησαν στο JCPA σε σχέση με την ε, συμφωνία αυτή, την συμφωνία με το Ιράν και βλέπουμε τι επιπτώσεις υπάρχουν από την αποχώρηση των ΗΠΑ. Είδαμε τα νομικά κείμενα, προσπαθήσαμε να κάνουμε μία σύνοψη και στο παράρτημα έχετε δύο διαφορετικές περιληπτικές αφορές. Καταρχάς, συμμόρφωση. Τι περιμένετε να μην γίνει, τι περιμένουν οι να μην κάνουν οι επαρκές σε σχέση με το Ιράν και δεύτερον, ε, η βλάβη στα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Τι μπορεί δηλαδή να επιβάλλει ως στις ε, μερικοί στους ε, ευρωπαϊκούς οικονομικούς φορείς. Εάν ε, προβούν σε ενέργειες που είπατε θα ήθελαν να προβούν. Αυτό λοιπόν σε μεγάλο βαθμό έγινε σε συνεργασία με την Επιτροπή FBI αλλά σε στενή συνεργασία με τους συναδέλφους από την ΕΙΕΔ και για την προσωπία των Ένωση στην που συμμετείχε σε, αυτή. την, σε αυτό το εγχείρημα. Θεωρούμε ότι ε, δεν είμαστε εκεί πλέον ειδικοί, οπότε καλό ήταν να μας βοηθήσει και αυτή η αντιπροσωπεία. Και το παράρτημα το είδαν ε, και Αμερικανοί δικηγόροι που είναι ειδικοί στα θέματα των κυρώσεων και θεωρούν ότι είναι καλά αυτά τα οποία περιλαμβάνει το παράρτημα. Άρα πιστεύουμε ότι έχουμε ένα καλό παράρτημα. Υπάρχουν αρκετές νομικές πράξεις ε, που περιλαμβάνονται στο παράδειγμα και ένα κανονισμός. Ε, έχουμε τον νόμο για τι κυρώσει στο Ιράν ε, που θεσπίζει και κυρώσει για τα πετρελοειδή, πετροχημικά, δράση για την ελευθερία και κατά τη διάδοση των όπλων, για το Ιράν, ενέργεια, κυρώσεις το μετσανίσεων και για τους εξωτερικού φορείς και και ο νόμος του 12 για τις ε, εξόδου ε, ε, National Defense Authorization για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη Συρία, για το δημόσιο χρέος. Και ο κανονισμός για τις συναλλαγές με το Ιράν για αγαθά και υπηρεσίες από τις είπα που δεν θα πρέπει να έπαν εξάγονται στην Ευρώπη. Υπάρχει πάγωμα πεσοκών στοιχείων, απαγόρευση πρόσβαση στις αγορές, αυτές οι νομικές πράξεις επίσης και υπάρχει για το 12 αυτό το National Authorization που σας είπα για χρηματικές και ποινικέ κυρώσεις. Πολύ σημαντικό θέμα. Δεν θα σας πω τι λέει ο κανονισμός παρεμπόδισης. Ουσιαστικά προστατεύει τους οικονομικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. για να μην υπάρξει αναγνώριση επιβολή στην Ευρωπαϊκή Κανενός από αυτό, αυτά τα νομοθετήματα που σας ανέφερα πριν και για να προστατευθούν από κυρώσεις οι εταιρείε μας. Υπάρχει επίση υποχρέωση ενημέρωση κομισιών για τον αντίκτυπο της νομοθεσίας στους οικονομικού μας φορείς. Αυτό θα είναι η βάση για εμάς ώστε να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο αυτών των κυρώσεων όταν ε, αρχίσουν να ισχύουν εκ νέου, ελπίζοντα να μα ενημερώσουν για τα αποτελέσματα αυτών οι οικονομικοί φορεί. Ε, Επιπροσθέτω όλα αυτά. Έχουμε εκτό του κανόνα παρεμπόδιση το διαρθρωμένο διάλογο με τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή. Γιατί τα κράτη-μέλη έχουν αρκετέ απορίε για το πώ θα εφαρμοστεί. Νομοθεσία δεν έχουν εμπειρία. Γιατί σα είπα, ο κανονισμό ήταν ουσιαστικά ανενεργός. Επίσης, υπάρχει ένα σοβαρός διάλογος με το Ιράν. Ε, με τους αδέλφους από την ΕΕ πήγαμε στη Τεχεράνη πρόσφατα, συζητήσαμε διάφορα θέματα που άπτονται των κυρώσεων και των οικονομικών ωφελιών. με το τμήμα των κυρώσεων κατά του Ιράν. Υπάρχει επίσης ε, πραγματικά ε, μια καλή συνεργασία με γάμα δέλτα εμπόριο, Move, ενέργεια, βίσμα για ε, την αντιμετώπιση της κατάστασης. Uh, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Καλύψατε όλη την κατάσταση αναφερόμενη και σε αυτές τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Δεν έγινε όμω αναφορά στην αναδιατύπωση, έτσι δεν είναι, στι διαφορετικέ συναλλακτικέ που υπήρχαν. Αναφέρθηκε σε αυτό η κυρία Μογκερίνη. Είπε ότι θα μπορούσαμε να διαρευνήσουμε άλλε συναλλακτικέ. Υπάρχουν εναλλακτικέ σε σχέση με την αναδιατύπωση ή όχι. Ναι, ναι, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Μα μακάρι να μπορούσα να σας φέρω χαρμόσυνα νέα, ότι δηλαδή τρεις νομικές υπηρεσίες κατέληξαν συμφωνία και ότι μπορούμε να συνεχίσουμε. Δυστυχώς δεν έχω τέτοια χαρμόσυνα νέα και όσον αφορά την, τις πιθανές ε, τροποποίησεις ε, στον κείμενο, πέρα από την αναδιατύπωση δηλαδή, το ζήτημα αυτό το λάβαμε ως ερώτηση από τα κράτη-μέλη και από τους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι είπαν ότι θα μπορούσε το κείμενο αυτό να γίνει λίγο πιο στιβαρό, αν θέλετε, να έχει μεγαλύτερη ισχύ. Δεν έχουμε αποκλείσει αυτή την εναλλακτική, απλώς αναφέρθηκα μόνο στις κατεξιότηση πράξεις διότι ε, Ήδη έχουμε κάπως καθυστερήσει. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι αυτές οι οποίες ε, έθεσαν, να θέλετε, το ρυθμό τη όλη διαδικασία, αποχωρώντας από τη συμφωνία. Επομένω, έπρεπε εμεί να αντιδράσουμε γρήγορα, πολύ γρήγορα, για να καθησυχάσουμε του οικονομικού φορεί στι αγορέ και προκειμένου να του προστατεύσουμε το καλύτερο δυνατό τρόπο. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο συζητήσαμε μόνο τον κανόνα παρεμπόδισης. Τώρα, μία τροποποίηση για τον κανονισμό, αυτός δεν έχει συζητηθεί ως πρόταση επίσημη, αλλά προφανώς να αποκλείεται αυτή τη στιγμή. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Ο κύριος Χέφνερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω εκ μέρους του γιατί είναι ο σκιώδης ε, του ΕΛΚΑ για αυτό το ζήτημα. αλλά δεν θα μιλήσω στα πολωνικά όπως Ο κύριος Λουμπανοβαρής λοιπόν, ευχαριστεί τον συγκεκριτή για αυτό το έγγραφο εργασία. Ε, και τρία σχόλια έχει να κάνει. Ε, καταρχήν πρόκειται για ένα έγγραφο που έρχεται στη σωστή χρονική συγκυρία, γιατί όλοι παρακολουθούμε τι διεθνεί εξελίξει και την απόφαση των ΗΠΑ να εγκαταλείψουν την συμφωνία, την κοινή ε, συμφωνία, ολοκληρωμένη συμφωνία για το Ιράν. Και βέβαια πρόκειται για μια ε, απόφαση που έχει λάβει η Αμερικανική πλευρά, ε, κυρίαρχη απόφαση, αλλά η οποία έχει επιπτώσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό θα πρέπει να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση. Το δεύτερο σχόλιο είναι ότι ε, πως αυτή η συμφωνία σε ό,τι αφορά τον κανόνα παρεμπόδιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάπως παροχημένη και, παροχημένη και χρησιμοποιεί δηλαδή μια ορολογία πριν από 20 χρόνια. Ε, άρα λοιπόν η ε, νομοθετική διαδικασία αφορούσε ειδικότερα τα ζητήματα σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Κούβας Ενώ με το Ιράν ε, το όλο ε, σύστημα και οι κυρώσεις έχουν διαφορετικό χαρακτήρα. Οπότε ένα τέτοιο σύστημα δεν μπορεί να είναι χρήσιμο ε, για αυτό το σκοπό και ο κ. Βαλένσα συμφωνεί με το ότι θα πρέπει να εξορθολογιστεί αν θέλετε εδώ το σύστημα. Αλλά το τρίτο σχόλιο του κ. Βαλένσα είναι κάτι το οποίο σχετίζεται και με το ερώτημα που έθεσε ο κ. Σελάγκη. Ότι δηλαδή εμ, διερωτάται για το γεγονός ότι αντί να προβεί σε επανεξέταση του όλου συστήματος και του παλιού κανονισμού προβαίνει σε, σε απλώς ένα recast, σε μία αναδιατύπωση. Γιατί ε, με μια τέτοια γενικότερη αναθεώρηση θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη μας το σημερινό σύστημα κυρώσεων. Ε, κάτι το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο. Οπότε, εσεί ήδη θέσατε πρόεδρε το ερώτημα, αλλά ο Σάντζο Βαλέζα ήθελε να θέσει ακριβώ αυτό το ερώτημα στην Επιτροπή. Ότι δηλαδή, γιατί αποφάσισε να προβεί σε μια αναδιατύπωση, σε ένα ρίκαστερ. Ε, καθώς περιορίζει τις δυνατότητες ε, που έχουμε σε ό,τι αφορά τα αναθεώρηση του συστήματος. Ε, ε πάντως, ο κ. Βαλέσσα ε, αναμένει με ενδιαφέρον τη συνεργασία που θα έχει με τον εισηγητή σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σάκη έχει το λόγο. Σημαντικό το ζήτημα αυτό, αλλά θα πρέπει να είμαστε και πάρα πολύ συγκεκριμένοι όσον αφορά τα νομικά και τα πολιτικά μέτρα, νομικά μέτρα και πολιτικές προκλήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να έχω περισσότερες πληροφορίες για αυτή την έννοια του κανόνα παρεμπόδισης που θα επέτρεπε τελικά τελικά από κάποιες εταιρείες να αποζημιωθούν, από τις χώρες εκείνες που έχουν επιβάλει κυρώσεις. Στην πράξη τι θα γίνει, ας πούμε ότι είστε μία τράπεζα, ότι έχετε επενδύσει εκατομμύρια και ότι ξαφνικά ζημιώνεστε πάρα πολύ σημαντικά. Σε ποιον θα απευθυνθείτε στην Αμερική, στη δική του την Κεντρική Τράπεζα, πώς ακριβώς θα γίνει και τι θα γίνει και με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Ερχόμενοι εσείς, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε επαφή με τον ιδιωτικό τομέα, με τις επιχειρήσεις, τι διδάγματα έχετε αποκομίσει. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που αναφέρθηκε σε διάφορα άρθρα στα μέσα ενημέρωση. Θεωρώ και εγώ ότι είναι σημαντικό να αποφύγουμε να αναλάβουν τα δημόσια θεσμικά όργανα ένα πολύ μεγάλο ιδιωτικό κίνδυνο. Θα είναι μη βιώσιμη η κατάσταση αυτή και θα οδηγήσει, αν θέλετε, σε λαθασμένα κίνητρα. Τώρα, από πολιτικής πλευράς, αν το Κογκρέσο και ο Πρόεδρος των Πολιτειών όντως έχουν την πρόθεση να αυξήσουν τις κυρώσεις εις βάρος του Ιράν, τότε υπάρχουν και πολλές άλλες διάβλοι ουσιαστικά που τους συνδέουν με το πρόγραμμα του Ιράν. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να είχαμε κυρώσει όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, κυρώσει όσον αφορά την πολιτική στάση του Ιράν στην περιοχή. Έχετε ασχοληθεί καθόλου με την πτυχή αυτή, αν υπάρχουν κυρώσει άλλη φύση και τότε πώς επηρεάζεται και το blocking status, ο κανόνας παρεμπόδισης. Ο κανόνας παρεμπόδισης έχει να κάνει μόνο με τις κυρώσεις που έχουν να κάνουν με το πυρηνικό πρόγραμμα ή γενικά συνδέεται με τα γενικότερα εξοδαφικά μέτρα τα οποία οι Ηνωμένε Πολιτείε μπορούν να λάβουν κατά του Ιράν και για πολλούς άλλους τομείς δηλαδή. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει στο ζήτημα αυτό να καταφέρουμε εμείς να ανταποκριθούμε πολύ δυναμικά για να μην χάσουμε την αξιοπιστία μας Βρισκόμαστε εν γέννη σε μια αμυντική αυτή τη στιγμή στάση όσον αφορά το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράση με το Ιράν. Θα πρέπει να εμείνουμε στάση, έχουμε υπογράψει, να παραμείνουμε μια αξιόπιστη δύναμη. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα ζητήματα από των οποίων έχουμε κάθε δικαίωμα και κάθε ευθύνη τελικά να είμαστε πολύ πιο σαφεί ω προ το πού βρίσκονται τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και οι ευρωπαϊκέ αξίε. και ας είμαστε προσεκτικοί τη γενικότερη εντύπωση που δίδεται από την όλη συζήτηση. Δεν θα πρέπει να φαίνεται ότι θέλουμε μόνο να προστατεύσουμε αυτό το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης με το Ιράν και ότι ε, συστρατευόμαστε τελικά με τη μία ή την άλλη δύναμη Αμερική ή Ιράν, θα πρέπει να φαίνεται από την όλη αυτή στάση και συζήτηση ότι προασπιζόμαστε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και τις ευρωπαϊκές αξίες. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ζαντό έχει το λόγο σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σάκε ήδη προχώρησε σε πολύ αυστηρά μέτρα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί αυτή τη στιγμή πίνει από ό,τι βλέπω μια κοκακόλα κολα χωρίς ζάχαρη και όχι μια κανονική κλασική κοκακόλα. Σε σχέση με αυτά που είπαν και οι συνάδελφοι, συμφωνώ και εγώ ότι το ζήτημα είναι σαφώς πολιτικό. Κοιτάξτε, για μένα το ότι η Total δεν μπορεί να πάει και να εξορίξει πετρέλαιο φυσικό αέριο στο Ιράν δεν είναι για μένα το πιο σημαντικό πρόβλημα. Ξέρετε ότι οτιδήποτε και να λέμε εμεί, ανεξάρτητα με το τι αποφασίζουμε, η Total και άλλοι μεγάλοι όμιλοι θα πάρουν τι αποφάσει του. Σε κάθε περίπτωση θα προτιμήσουν να έχουν καλέ σχέσει με τις ΗΠΑ από ότι με το Ιράν. Αυτό είναι σίγουρο. Το ζήτημα τέθη μάλιστα πολλέ φορέ. Τι θα γίνει στην πράξη. Για παράδειγμα, για μια μικρομεσαία ευρωπαϊκή επιχείρηση, η οποία λόγω της συνδίκευσής της δραστηριοποιείται στην αγορά του Ιράν. Τι θα γίνει με μια τέτοια επιχείρηση. Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θα ζητήσουν, ε, για παράδειγμα, να κατασχεθεί το Air Force One αυτή τη στιγμή πατήσει σε ευρωπαϊκό έδαφος ή θα προχωρήσουν σε άλλα μέτρα. Όπως και άλλοι συνάδελφοι δεν κατάλαβα τελικά πολύ καλά πως στην πράξη θα οργανωθεί η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς ευρωπαϊκές εκείνες επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να παραμείνουν στο Ιράν διότι τελικά οι οικονομικές προοπτικές εκεί πέρα είναι πολύ πιο πολλά υποσχόμενες από τις Ηνωμένες και όπως και οι συνάδελφοι, και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η στάση μας. Δεν βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην περίπτωση της Κούβας, ούτε διανύουμε την περίοδο Κλίντον, διανύουμε την περίοδο της προεδρίας του Τραμπ και θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να προσαρμοστεί και δική μας η στάση. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κάμπελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξέρω ότι α, αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για εξωτερικές υποθέσεις στην Επιτροπή μας, δεν είναι η άμεση αρμοδιότητά μας. Αποφασίσαμε να μην προχωρήσουμε σε εμπορική συμφωνία με την Κίνα λόγω των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και τώρα μιλάμε για εμπορική συμφωνία, εμπορικέ δραστηριότητε με το Ιράν, που ξέρω ότι έχει το χειρότερο ρεκόρ εκτελέσεων στον κόσμο. Σήμερα το πρωί διάβαζα ένα άρθρο για μια εκτέλεση που έγινε χθε στο Ιράν. Ένα άνθρωπο του οποίου του σπάσανε τα δόντια, τον χτύπησαν, τον ξυλοκόπησαν, χρειάστηκε να κάνει ράματα, χρειάστηκε να υπογράψει εν συνεχεία, ο Μοχάμετ Σάλε ονομάζεται, μια ψευδή δήλωση και εν τέλει ο άνθρωπο αυτό μετά από όλα αυτά τα βασανιστήρια εκτελέστηκε χθε. Για ποιο λόγο συνεργαζόμαστε με το Ιράν, έχουν δίκιο οι ΗΠΑ, κάνουμε ένα τεράστιο λάθο, δεν πρόκειται να πετύχουμε τίποτα απολύτω. Ξέρετε ότι κάνανε ε, δοκιμές βαλιστικών πυράβλων έχουν αποσταθροποιήσει εντελώ την ε, Μέση Ανατολή και πρέπει να σας πω ότι ε, αυτή τη στιγμή οι κυβερνώντες στο Ιράν αποσταθροποιούν και την ίδια τη χώρα οι φράξεις οι οποίες συμμετέχουν στην κυβέρνηση του Ιράν. Και εμείς τροφοδοτούμε και ενισχύουμε την κυβέρνηση αυτή και αυτό το καθεστώς μέσω του εμπορίου. Θεωρώ λοιπόν το ζήτημα είναι σαφώς περισσότερο πολιτικό και ζήτημα εξωτερικών υποθέσεων από ότι εμπορικό. Είναι πραγματικά επονίδιστο αυτή τη στιγμή το ότι εμπορευόμαστε με το Ιράν και ότι έχουμε αποκλείσει την Κίνα. Είναι πραγματικά πρόδειλη και επονίδιστη η ασυνέπεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε όλες αυτές τις ιδεχθείς εκτελέσεις οι οποίες σε καθημερινή βάση συνεχίζονται στο Ιράν. Σας ευχαριστώ. Αυτό είναι ένα από τα λίγα πράγματα για τα οποία δεν έχω άποψη γιατί δεν γνωρίζω πολλά για αυτό το άκρο τεχνικό ζήτημα. Είναι εντυπωσιακό όμω που η Ισραηλινή κυβέρνηση που έχει αυτή την υπηρεσία πληροφοριών συστηματικά είναι αντίθετη και ήταν αντίθετη πάντοτε σε αυτή, την αρχική, ε, σε αυτή τη συμφωνία. Έχω ένα τεχνικό ερώτημα προς την ε, Κομισιόν. Όσοι έχει κατάσταση αυτή τη στιγμή, Μα δώσετε μια πολύ αδρή, ε, μπορώ να σας κάνω μια πολύ αδρή σύνοψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Μάλλον όχι. Οι Ηνωμένε Πολιτείε αποσύρθηκαν, αποχώρησαν από τη συμφωνία και επιβάλλουν Ρώσοι στο Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το κάνει. Εντάξει, παραπλουστευμένα σας τα λέω, ίσως απλοϊκά, αλλά ε, αυτό είναι ουσιαστικά. Ιδίω ε, στον οικονομικό τύπο λέγεται ότι επειδή είπα ελέγχουν το σύστημα καθάρισης ε, ό,τι κι αν κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν οι επιβάλλουν ε, κυρώσεις και για όσο το κάνουν αυτό θα υπερτερούν λόγω αυτού του συστήματος Πέλε. Θα ήθελα να μας ενημερώσει η Κομισιόν για το κατά πόσο αυτό που είπα είναι αληθές ή ψευδές. Κύριος Ρούμπιχ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή γιατί εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με το Ιράν, αλλά με τη γενική αρχή του πώς θα πρέπει να αντιδρούμε όταν επιβάλλονται κυρώσεις ε, από εταίρους με τις οποίες εμείς δεν συμφωνούμε. Ε, αναφερθήκαμε εδώ βέβαια στις δυνατότητες ε, παρεμπόδισης που έχουμε εδώ, τα blocking options, αλλά ε, το ερώτημα που τίθεται είναι τι θα πρέπει να κάνουμε στις ε, αντίθετες περιπτώσεις. Δηλαδή όταν ε, δεν θέλουμε να προβούμε σε παρεμπόδιση, αλλά θέλουμε ακριβώς να επιτρέψουμε κάποιες εμπορικές συναλλαγές. Ιδιαίτερα για παράδειγμα στον χώρο της ενέργειας θα ήταν χρήσιμο να εξετάσουμε το κατά πόσο στο μέλλον θα έπρεπε να γίνονται οι σχετικέ συναλλαγέ μέσω ευρωπαϊκών συναλλαγών. Νομίζω πω και τα δύο νομισματικά συστήματα βρίσκονται ε, σε ανταγωνισμό και ως το Ιράν μέσω ε, του ΟΠΕΚ έχει αναλάβει κάποιε δεσμεύσει. Όμω ε, από την άλλη πλευρά με την Ευρωπαϊκή Χάρτα θα πρέπει να εξασφαλιστεί και η αμοιβαιότητα. Άρα λοιπόν πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε την αμοιβαιότητα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ε, της Ενεργειακής ε, Χάρτας έτσι ώστε να βρεθεί σε μια ισχυρή θέση Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Αμπεκίνη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και εγώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους εμπειρογνώμονες για τις παρεμβάσεις τους. Εγώ βλέπω ευνοϊκά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, σε σχέση με την τροποποίηση του κανονισμού αυτού που έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των κυρώσεων κατά του Ιράν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό χάρη στη δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μπορούν ε, να προστατεύονται οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από την εξοδαφική εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνουν οι ΗΠΑ. Οι κυρώσει αυτές ακούσαμε ότι θα επιβληθούν σε δύο στάδια, τον Αύγουστο και τον Νοέμβριο και θεωρώ ότι θα πρέπει μέσω του δικού, μου, δικού μας του κανονισμού να προστατεύσουμε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Έχω κάποιε αμφιβολίες, θα ήθελα να τι διασκεδάσει η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφέρομαι σε μια ευρωπαϊκή επιχείρηση η οποία ενδεχομένω να έχει επενδύσει στο Ιράν και να πλήττεται τώρα από τι κυρώσει ε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την επιχείρηση αυτή. Γιατί ξέρετε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε βασικά ε, δεν θα επιτρέψουν σε αυτή την επιχείρηση να λειτουργήσει φυσιολογικά και θα χάσει ουσιαστικά πάρα πολλά κέρδη. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι υπάρχουν προστευτικά μέτρα στον κανονισμό. Ποιο ακριβώ όμω θα αποζημιώσει την επιχείρηση αυτή που θα ζημιωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αρμόδιες αρχέ των ΗΠΑ που έχουν επιβάλει εξοδαφικά τα μέτρα αυτά. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι ΗΠΑ να λάβουν ένα μεγάλο βάρο τη αποζημίωση αυτή. Επίση, είναι πάρα πολύ σημαντικό όλα τα κράτη-μέλη με τον ίδιο τρόπο να εφαρμόζουν τα αντιμέτρα, προκειμένου να μπορέσει ο κανονισμό αυτό ομοιόμορφα να ισχύσει. Ευχαριστώ. A lot of questions. Ωραία, πολλά ερωτήματα. Να δώσω λοιπόν καταρχήν ε, πρώτο λόγο στον κύριο Ντεβιδιά Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πως τα περισσότερα από που θέθηκαν ε, απευθύνονται προς την Επιτροπή. Ε, και έχουμε πάντως εδώ μαζί μας το συνάδελφο από την Task Force για το Ιράν που ενδεχομένω θα ήθελα να πάρει το λόγο. Πάντως επιτρέψτε μου εγώ να κάνω ένα σχόλιο σε ό,τι αφορά την ε, γενική συμφωνία ε, με το Ιράν και τις δράσεις του Ιράν για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και την εμπλοκή του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή. Νομίζω πως η συμφωνία αυτή έχει ένα και μόνο στόχο και αυτό είναι να παρεμποδίσει τη χρήση ε, πυρηνικών όπλων από την πλευρά του. Δεν είναι ο στόχο τη συμφωνία να επιλύσει ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπάρξει πολύ ξεκάθαρη και σαφή ω προ τη στάση τη απέναντι σε αυτά τα ζητήματα ε, και ήδη έχουμε εφαρμόσει κυρώσει σχετικέ ε, σε ό,τι αφορά ανθρώπινα δικαιώματα ε, για 82 συγκεκριμένα άτομα. Έχουμε από εκεί και μετά κάποιες ακυρώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την ε, διάδοση όπλων και σχετίζονται και με την Γενική Συμφωνία. Έχουμε από εκεί και μετά ε, κυρώσεις που έχουμε επιβάλει στο Ιράν σε ό,τι αφορά τη στάση της απέναντι στη Συρία, αλλά και κυρώσεις που αφορούν την ε, υποστήριξη της τρομοκρατίας από την πλευρά αυτής της χώρας. Αυτά λοιπόν όλα εντάσσονται στη γενική μας ε, προσέγγιση εδώ ε, και δεν ξέρω αν επιτρέπετε Πρόεδρε ο κύριος Τσαβγέ μετά από τη συνάδελφο από την Επιτροπή να πάρει το λόγο και να κάνει και εκείνο κάποια σχόλια. Καλώς λέει ο Πρόεδρος Λάγκη. Επιτροπή λοιπόν. Σας ευχαριστώ για αυτά τα ερωτήματα. Θα προσπαθήσω να τα ομαδοποιήσω, παρότι δεν είχα πολύ καιρό στη διάθεσή μου για να το κάνω. Ξεκινώ λοιπόν με το πρώτο ερώτημα, ως προς το γιατί επιλέξαμε να προβούμε σε ένα recast, σε μια διατύπωση του κανονισμού. Αν αναφέρεστε σε εκείνο το recast του 2015 και τη σχετική πρόταση, ε, τότε είχε προταθεί ένα, ε, μια τεχνική, τεχνικού χαρακτήρα βελτίωση Οπότε ε, τα πράγματα έχουν αλλάξει αυτή τη στιγμή και ε, βέβαια είπαμε ότι θέλαμε κατεξοδότηση πράξη ώστε να υπάρξει μια ταχεία λύση για να δώσουμε και το κατάλληλο σήμα ε, στις αγορές μας και στους εμπορευόμενους μας αλλά να δώσουμε ταυτόχρονα και ένα πολιτικό μένουμε προς το ΕΡΑΝ. Τώρα, το ζήτημα που μας αφορά σε ό,τι αφορά τον κανόνα παρεμπόδισης και το κατά πόσο αυτό είναι μόνο το, η χρήση πυρηνικών όπλων ή όχι, η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, τότε όταν είχε εφαρμοστεί ο συγκεκριμένο κανονισμό δεν αφορούσε καν, δεν είχε προκύψει καν αυτό το πυρηνικό ζήτημα και αφορούσε στην προστασία γενικότερα τη Ευρωπαϊκή Ένωση από τέτοια μονομερή μέτρα. Ε, τώρα λοιπόν έχουμε το ΕΡΑΝ στο παράδειγμα, αλλά δεν υπάρχουν περιορισμοί στο τι μπορεί να καλύψει ο κανονισμό. Πάντω με αυτή την βελτίωση στην οποία προβαίνουμε τώρα είναι ακριβώ η κάλυψη αυτή τη περίπτωση όπου έχουμε επιβολή μονομερών μέτρων από τις Πολιτείες απέναντι στο Ιράν. Τώρα, και τώρα η πιο σημαντική ερώτηση από όλες είναι το πώς ε, γίνεται η ανάκτηση αν θέλετε αυτών των ζημιών και ε, πραγματικά είναι μια θεμητή ερώτηση την οποία έχετε θέσει και θα ήταν ψέματα του να σας πω ότι έχω μία απόλυτη απάντηση. Γι' αυτό προφανώς ε, δεν αποτελεί πανάκια ένας τέτοιος κανονισμός. Ε, δεν θα επιλύσει όλα τα προβλήματα. Και αυτό ε, το λέω και απαντώντας στα σχόλια τα οποία έγιναν σε ό,τι αφορά την ε, προνομιακή αν θέλετε ε, θέση του Ευρωπαϊκού, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, γιατί ναι μεν έχουμε προνομιακή θέση αλλά οι Ηνωμένες έχουν πολύ μεγαλύτερη ισχύ στην παγκοσμιωμένη οικονομία. Αυτό όμως προσπαθούμε να κάνουμε με τους αυτούς τους κανόνες παρεμπόδισης και ειδικότερα με την διάταξη σε ό,τι αφορά την ανάκτηση των ζημιών είναι να διαβεβαιώσουμε τις επιχειρήσεις ότι παρόλες τις απειλές ε, και τις επιθέσεις είμαστε διατεθειμένοι να έρθουμε σε επαφή με το Ιράν, να συζητήσουμε και να ανακτήσουμε τις ζημίες αυτές. Και το πώς μπορεί να γίνει ανάκτηση δεν είναι μια, ένα ερώτημα το οποίο μπορεί να απαντηθεί με ένα ναι ή με ένα όχι. Ε, σε ό,τι αφορά το επίπεδο ε, και το από ποιον γίνεται η ανάκτηση, εδώ βρισκόμαστε και στον, στην σύμβαση των Βρυξελών, ε, δηλαδή ε, δικαστικά από τον αρμόδιο φορέα και η διαδικασία αυτή, η δικαιοδοσία για την διαδικασία αυτή αφορά το δικαστήριο ε, στο οποίο έχει την έδρα του επιχείρηση το άτομο το οποίο έχει υποβληθεί έχει υποστεί τη ζημία έτσι ώστε να μπορέσει να ανακτήσει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Οπότε δεν μπορώ να σας δώσω μια πιο ξεκάθαρη απάντηση γιατί ε, θα εξαρτηθεί από την ομοθεσία του εκάστοτε αρμόδιου δικαστηρίου η το πώς ακριβώς θα γίνει η προσφυγή και πώς θα γίνει η ανάκτηση των σχετικών στοιχείων από την άλλη πλευρά. Τι άλλο έχω σημειώσει τώρα εδώ από ερωτήσεις. Ναι, νομίζω πως τα κάλυψα όλα ε, και σε ό,τι αφορά την προνομιακή θέση των Ηνωμένων Πολιτειών, σε ό,τι αφορά τις χρηματοοικονομικές αγορές. Όπως είπα, ναι, το γνωρίζουμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ε, περκεράσουμε αν θέλετε αυτή τη δυσκολία και προκειμένου να ε, ε, διασφαλίσουμε την οικονομική μας κυριαρχία, αν θέλετε, παρά αυτήν την κυρίαρχη θέση των ΗΠΑ. Επίσης, αναφέρθηκε και αυτή η πρόταση ενός πακέτου με μέτρα που δίνουν περαιτέρω δυνατότητε σε συναλλαγών, enabling, αν θέλετε, και όχι μόνο διατάξει σε ό,τι αφορά παρεμπόδιση. Πράγματι, έχουμε ξεκινήσει αυτή την εξέταση και υπάρχουν μια σειρά από γενικέ διευθύνσει που έχουν εμπλακεί σε αυτή τη συζήτηση ω προ το ότι δηλαδή όχι μόνο να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να αμυνθούν από τις ε, μονομερεί ε, κυρώσει από την πλευρά των Πολιτείων αλλά και προκειμένου να υπάρξουν περαιτέρω διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά τι συναλλαγέ του ε, με το Ιράν. Και υπάρχουν εδώ παραδείγματα από διάφορου τομεί τη οικονομία, για παράδειγμα ενέργειε, μεταφορά, ασφαλίσει Εξετάζουμε λοιπόν αυτά τα ε, στοιχεία και φυσικά χρειαζόμαστε και κάποιο χρόνο. Γιατί σε ορισμένε περιπτώσει βέβαια είναι δυσκολότερο το να προωθήσουμε ακριβώ ε, να διευκολύνουμε τέτοιου είδου από το να μπλοκάρουμε αρνητικέ ε, κυρώσει. Ευχαριστώ, λέει. Πρόεδρο Μόνικα, θέλει να προσθέσει τίποτα. Να προσθέσω και εγώ κάτι σε σχέση με την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων αυτών που συνεχίζουν και επενδύουν ε, στο Ιράν. Ακούσαμε ότι υπάρχουν ορισμένε επιχειρήσει που ενδεχομένω να αποσυρθούν. Όσον αφορά πιο συγκεκριμένα τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, δεν αναφέρομαι εδώ πέρα βέβαια μόνο στι μικρέ επιχειρήσει αλλά και τι μεσαίες επιχειρήσει και ξέρω ότι πολλέ τέτοιε επιχειρήσει είναι ευρωπαϊκές. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια όπω σα είπα προκειμένου να συνεργαστούμε με το Ιράν μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στις δύο πλευρές. Και προτού δούμε αυτές τις τελευταίες εξελίξεις, ακόμα και για το χρηματοπιστωτικό τομέα, βλέπαμε ότι ήταν οι μικρότερες ευρωπαϊκές τράπεζες εκείνες οι οποίες δεσμευόντουσαν με την Ιρανική οικονομία και που μπορούσαν να λειτουργήσουν στα πλαίσια του Ιράν. Είμαστε λοιπόν σε επαφή με την Ιρανική κυβέρνηση και συζητάμε και με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έχετε το λόγο. Θα ομαδοποιήσω σε δύο κατηγορίες τις απαντήσεις. Πρώτη, η ομάδα σχέσεις ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιράν και δεύτερο, οικονομικά κίνητρα και ΜΜΕ. Λοιπόν, για τις σχέσεις ε, Ιράν-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έγινε αναφορά σε μια υπόθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την γνωρίζω και ο πρόσωπος ε, του HRVP έκανε χθε μια σχετική ανακοίνωση με τις συζητήσεις που έχουμε για το ε, Ιράν, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε ένα διάβλο επικοινωνία που είναι θετικός, χωρίς ε, να ε, επικυρώνει ότι γίνεται οτιδήποτε, προσπαθεί να αλλάξει κάπως την κατάσταση. Για να σα δώσω ένα παράδειγμα, είχαμε επικοδομητική συζήτηση με το Ιράν για την ε, θανατική ποινή ε, σε αυτού που υποπέμπουν σε παρά το σχετικό με τα ναρκωτικά. Και είχαμε μεγάλη μείωση του αριθμού εκτελέσεων σχετικά. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Όμως όποτε έχουμε τις αντίστοιχες με τη χθεσινή καταστάσεις, αυτό που κάνουμε είναι ότι τηλεφωνούμε και προσπαθούμε με οποιοδήποτε τρόπο να παρέμβουμε. Σε ό,τι αφορά το αν οι ΠΑ έχουν δίκιο ή όχι, που αποχώρησαν από τη συμφωνία. Πάκτα sunt σερβάντα Αν υπάρχουν κανόνες και έπειτα δύο χρόνια μετά κάποιος ε, επαναχωρεί, αυτό δεν οδηγεί σε ένα σταθερό κλίμα και σε σταθερές σχέσεις. Άρα δεν είναι το θέμα ποιος έχει δίκιο και ποιος δεν έχει, αλλά να δούμε ποιος είναι ο κίνδυνος σε μια πολύ ρευστή ασταθή περιοχή, που υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες έχουν ε, τεράστιες ε, δυνατότητες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για καταστροφικούς σκοπούς. Και Αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμεί είναι να προφορτήσουμε την κατάσταση και όχι να δούμε ποιο έχει δίκιο ή άδικο, να βρούμε μακροπρόθεσμες λύσεις. αυτό είναι ο στόχος. Ε, και σε ό,τι αφορά το εμπόριο, 0,5 είναι η συναλλαγές μα με το Ιράν, αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, έχουμε σε ισχύ κυρώσει και γι' αυτό έχουμε αυστηρές ε, ε, διαδικασίες δέωσας επιμέλεια. Η σύγκριση με την Κίνα που είναι πάνω από 0,5% το όγκος των εμπορικών συναλλαγών ε, δεν είναι ξεκάθαρη. Και έρχομαι στα κίνητρα με τη δεύτερη επιμέλεια που σας προανέφερα. Κίνητρα μπορούμε να δώσουμε στους ευρωπαϊκούς οικονομικούς φορείς. Όπως είπαμε, έχουμε ε, το κανόνα παρεμπόδισης που στέλνει σαφή μηνύματα στους οικονομικούς φορείς ότι λειτουργούν σε ένα νόμιμο περιβάλλον, το περιβάλλον της Ένωση που δεν ε, υπόκειται σε κυρώσεις. Δεύτερον, η ΜΜΕ που είναι λιγότερο εκτεθειμένες από τις ε, πολυεθνικές έχουν μεγαλύτερη ευθεία κινήσεων ε, για να ε, συνάψουν κάποια οικονομική σχέση με το Ιράν. Αλλά θέλουμε να δούμε με τη δέωση επιμέλεια τι γίνεται με το καθεστώ και υπάρχουν και κάποιε άλλε δραστηριότητε και ενέργειε που μπορούμε να αναλάβουμε, τεχνική βοήθεια και διασκέψει που οργανώνουμε για τη ΜΜΕ για να καταλάβουν τι θα πει δέωση επιμέλεια και για να του παράσουμε τη σχετική υποστήριξη. Επίσης παρέχουμε τεχνική βοήθεια με, σε ιρανικές ΜΜΕ σχέσεις με την Ευρώπη για να καταλάβουν λίγο καλύτερα πώς λειτουργεί η ευρωπαϊκή αγορά ιδίως στον τομέα των τροφίμων και γεωργοδιατροφικών προϊόντων. Τέλος, κάτι πολύ σημαντικό που αναφέρατε για το βάρος τη βαρύτητα ε, των ΗΠΑ στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Πράγματι ισχύει αυτό ε, και αυτό συνιστά μεγάλη πρόκληση για να συνεχιστούν οικονομικέ ώρε μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ιράν. Ε, και να ζητούμε ιδιαίτερε λύσει, συγκεκριμένε λύσει, ε, που θα στέλνουν και ένα μήνυμα ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη ε, και διατεθειμένη να έχει τις δικές της, τους δικούς της οικονομικούς διάβλους. Θέλω επίσης να πω ότι το Ιράν αποφάσισε όλες τις εξαγωγές και συναλλαγές που κάνει σε πετρελαιοειδή να τις κάνει σε ευρώ. Και αυτό νομίζω ότι είναι θετικό για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε κάτι να προσθέσετε μήπως ε, κύριε Ζαντό. Εμείς είμαστε ε, εκλεγμένοι και μπορεί να μην είμαστε τόσο έξυπνοι ίσως, αλλά δεν ξέρω. Ε, έρχεστε εδώ, στην Επιτροπή μας και μας λέτε δώστε μας τη δύναμη να δράσουμε, γιατί πρέπει να είμαστε γρήγοροι. Όταν όμως σας ρωτάμε εμείς Πώ θα λειτουργήσουν όλα αυτά δεν έχετε να μα δώσετε κάποια σαφή απάντηση. Κατάλαβα ότι υπάρχει μια δέσμευση ε, να προστατεύσετε τι επιχειρήσει. Πόσο όμω θα το κάνετε δεν μα λέτε. Υπάρχει λοιπόν για μα και κάποια αντίφαση σε αυτή τη συζήτηση. Κύριε Σαλαφράγκα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στο ίδιο μικρό με τον προελίσσατε συνάδελφο. Έχουμε την πυρηνική συμφωνία από τη μία πλευρά, το Ιράν Προφανώ και έχει αναστείλει, απενεργοποιήσει τα δύο τρίτα των φοροκεντριτών και έχει φύγει αρκετά μεγάλη ποσότητα εμπεπισμένου ουρανίου από τη χώρα και επίσης οι δραστηριότητες των πυρικών έχουν ανασταλεί αποφάσισε με κυρίαρχη απόφαση τώρα η Αμερική να επαναθεσπίσει κυρώσεις αποχωρώντας από τη συμφωνία. Μας τα είπαν οι εκπρόσωποι τη ΕΕΔ. Οι κυρώσεις για το κεφάλαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, εν μέρει λειτουργούν. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς πρέπει την οικονομική μας κυριαρχία να επιβεβαιώσουμε και αυτούς τους ε, νόμους περί εξοδαφικής ε, εφαρμογής όπως ε, Helms Barton ε, δεν πρέπει να ε, έχουν αντικές επιπτώσει. δεν θα πρέπει να ισχύουν όπως και ο τελευταίος νόμος. Έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα όμως, έλλειψη εμπιστοσύνης. Καλό είναι να προσπαθούμε να προστατεύσουμε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, όμως φοβούμε Λαμβάνοντας δε υπόψη ε, ότι θα χαθεί ένα σημαντικό ε, ένα σημαντικό κομμάτι της αγοράς των ΙΠΑ δηλαδή. Οι δικές μας προσπάθειες πρέπει να εστιάσουν στην εξαίρεση από τις ΙΠΑ. Με βάση το τελευταίο σημείο, πακτάσουν τη Σερβάντα είπατε κι εσείς. Μετά από αυτά που μας είπε το πρωί ο Γενικός Διευθυντής για, για τα ζητήματα του εμπορίου, για το χάλιβα και το αλουμίνιο, Υπό τις συνθήκες αυτές θεωρώ αδύνατο να μπορέσει να ε, κερδίσει η εξαίρεση η Κομισιόν για τις Επιχειρήσεις ε, που ε, υπό την ομπρέλα της Πυρηνικής Συμφωνίας και επιμένω για πολιτικούς λόγους πρέπει να συμμετέχουν στις οικονομικές δραστηριότητες. Είναι πολύπλοκο πρέπει να επανεπιβεβαιώσουμε την οικονομική μα κυριαρχία, αλλά πολύ δύσκολα νομίζω ότι θα αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεών μας, που όπως είπα θα χάσουν ε, τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται στη σημαντική αυτή αγορά, τον είπα. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο για μια ακόμη φορά στην Κομισιόν, για... από τη δική μου πλευρά, φυσικά ίσως έχουμε και κάποιο αντίκτυπο ε, αυτό των εξωδικαστών εξοεδαφικών μέτρων τρίτων χωρών. Σε άλλε περιπτώσει. Έχουμε τη Ρωσία. Οι ΙΠΑ επιβάλλουν και, στις, ε, και στη Ρωσία ε, κυρώσεις. Αυτό ε, επηρεάζει και τι ευρωπαϊκέ εταιρείε. Θα υπάρξει και για αυτό το θέμα κάτι εξοδότηση πράξη. Feel θέλει το λόγο, διαλέξτε Ποιο θα ξεκινήσει. Ευχαριστώ. προσπάθησα, αλλά θα ξαναπροσπαθήσω να τα πω στο λεπτό πιο ξεκάθαρα, χωρίς να σας δώσω όμως και απαντήσεις ε, που δεν είναι τεκμηριωμένες. Πώς λειτουργεί ο κανόνας παρεμπό. Τρία προστατευτικά μέτρα. Ε, αποζημίωση, δυνατότητα αποζημίωση. Δεύτερο, αίτηση αδειοδότηση έγκριση από την Κομισιόν σε περίπτωση σοβαρή κινδύνου ε, στα συμφέροντα μιας επιχείρησης αν παραγνωρίσει ε, τις κυρώσεις ε, τον είπα, μπορεί να ζητηθεί αυτή η άδεια, αυτή η εξοδότηση, αν θεωρήσουμε ότι είναι αθέμητη η εξοδαφική εφαρμογή. Και τρίτη δυνατότητα, τρίτο προστατευτικό μέτρο δηλαδή, καμία απόφαση που θα βασίζεται σε εξοδαφικές αποφάσεις δεν μπορεί να επιβληθεί και να εφαρμοστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τελευταίο είναι σαφές. Κοινή απόφαση ε, από τη ΣΥΠΑ που λέει 2 εκατομμύρια πρόστιμο πληρώστε. Εμείς ε, θα πούμε, μάλλον οι θα πούν δεν γίνεται, δεν μπορεί να υπάρξει δίμευση, κατάσχεση περισσοκών στοιχείων. Αυτό είναι σαφές. Τι γίνεται με το σύστημα αυτό της αδειοδότησης. Δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει ή της έγκρισης, δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει. Τώρα καταρτίζουμε τα κριτήρια βάσει των οποίων μπορεί να δώσει αυτές τις άδειες η της εγκρισης δεν ξερουμε πως θα λειτουργησει τωρα καταρτιζουμε τα κριτηρια βασει των οποιων μπορει να δωσει αυτή τις αδειες η κομισιον και θα τα δούμε με την Επιτροπή για την εξεδαφική ε, νομοθεσία και ρύθμιση. Για να δούμε πώς εφαρμόζεται αυτό στην πράξη, γιατί δεν έχει γίνει κατά το παρελθόν. Δεν μπορώ να σας δώσω λοιπόν παραδείγματα, γιατί θα σας παραπλανήσω, θα σας ξαπατήσω. Για τις αποζημιώσεις όμως εδώ έχουμε κάποιο πρόβλημα. Σας έδωσα ήδη ένα παράδειγμα, μάλλον, ε, ναι, σε μια άλλη παρέμβαση. Πώς θα πληρώσω αποζημίωση, αν γίνει τότε δεν το δίνα. Πώς μπορούμε να το ξέρουμε είναι σαν να ε, λέμε αν κάποιος ε, ε, έχει ένα τροχαίο με πέντε οχήματα και ένα ζώο και ένα κόκκινο φανάρι, ποιος θα πληρώσει τα αποζημίωση. Α, τα κριτήρια αυτά υπάρχουν, αλλά τα δικαστήρια είναι αυτά που θα αποφασίσουν. Δεν μπορούμε εμείς να πούμε ως Κομισιόν τι θα αποφασίσουν τα δικαστήρια. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να είμαστε πιο ξεκάθαροι. Έχει να κάνει με την πρακτική εφαρμογή. Και αυτό θα είναι κατά περίπτωση. Σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Όταν υπάρχει ζημία για ευρωπαϊκή επιχείρηση. Αυτά είναι τα τρία βασικά. Αυτές είναι τρεις βασικές επιλογές. Και όπως είπα και στην πρώτη μου παρέμβαση, οι οικονομικοί φορεί βέβαια ίσως πρέπει να υποχρεωθούν να ενημερώσουν την Κομισιόν όταν έχουν πληγεί από την εφαρμογή ε, των εξεδαφικών αυτών νόμων, ε, όταν έχουν κυρώσει κτλ. Ε, γιατί εμεί, αν δεν ενημερωνόμαστε δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι αντίκτυπο έχουν, αν έχουν αυτέ οι κυρώσει. Από τη στιγμή που θα έχουμε αυτές τις πληροφορίε. θα μπορώ να σα δώσω και μια σαφέστερη απάντηση προ το παρόν. Δεν μπορώ να είμαι πιο σαφή. Ευχαριστώ. Uh, Σας ευχαριστώ. Να θίξω δύο σημεία όσον αφορά το ερώτημα για τη Ρωσία. Αν κατάλαβα καλά, μας ρωτήσατε αν θα επεκτείνουμε την επικαιροποίηση αυτού του κειμένου για να καλύψουμε και την Αμερικανική νομοθεσία σε σχέση με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες για πιθα νία εξοδαφική εφαρμογή ορισμένων μέτρων, ιδίως ε, των μέτρων εκείνων που προβλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ε, ως αντίπεινα σε κάποιες άλλες κυρώσεις. Ε, συζητάμε για όλα τα θέματα βέβαια με τις Ηνωμένες και συζητήσαμε και το ζήτημα των κυρώσεων επί της Ρωσίας και θα θέλαμε εκεί πέρα να αποφύγουμε τις ανεπιθύμητες συνέπειες των δράσεων αυτών, δηλαδή θέλουμε να αποφύγουμε τα αμερικανικά μέτρα κατά της Ρωσίας να έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε ευρωπαϊκές οντότητες, σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Συνεχίζει τη συζήτηση. αυτή, δεν από το τμήμα του blocking status, του κανόνα παρεμπόδισης, όσον αφορά το Ιράν. Συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και στο μέλλον όσον αφορά το ζήτημα των εξαιρέσεων, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να εφαρμόσουν τις κυρώσεις τους. Είναι ακόμα σαφές για μας σε πάρα πολλέ πτυχές τελικά πώ θα κινηθούν στο μέλλον. Δημοσίευσαν ένα κείμενο με ερωταπαντήσεις, με τις πιο συχνές ουσιαστικά ερωτήσεις και τις απαντήσεις που δίνουν οι ΗΠΑ. Συνεχίζουμε πάντως και συζητάμε μαζί τους για να δούμε πώς θα εφαρμοστούν οι κυρώσεις και αν θα υπάρχουν και πώς θα εφαρμοστούν κάποιες εξαιρέσεις. Και βέβαια αυτό δεν αποδυναμώνει σε καμία περίπτωση τη δική μας την ανεξάρτηση εντελώς τάση στα πλαίσια του κοινού αυτού ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για το Ιράν. Μία ακόμα ερώτηση θέλατε, έτσι δεν είναι. Ναι, μία ερώτηση τεχνική φύση. Έχουμε δύο εκπροσωπού από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Νόμιζα ότι στα μέλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μου λένε τώρα ότι δεν είστε. Έχουμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τρει εμπειρογνώμονε έχουμε. Έθεσα ένα τεχνικό ερώτημα, εσείς το παρακάμψετε, το αποφύγατε. Οι πολιτικοί δίνανται και μπορούν να αποφεύγουν έξυπνα τεχνικά ερωτήματα, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε το σύστημα του δολαρίου όσον αφορά την Παγκόσμια Τράπεζα. Το δολάριο χρησιμοποιείται για το παγκόσμιο εμπόριο πάρα πολύ και έχει γραφεί στον οικονομικό τύπο ότι σε σχέση με τις κυρώσεις αυτές εναντίον του Ιράν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να βγάλει ορισμένες τράπεζες από το σύστημα εκαθάρισης το οποίο βασίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο στο δολάριο. Έτσι λοιπόν οτιδήποτε και αν κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, λένε δημοσιογράφοι, ακριβώς επειδή οι Ηνωμένε Πολιτείε διατηρούν την απειλή τους αυτή στο παγκόσμιο σύστημα εκαθάρισης, ουσιαστικά πάντα θα υπερτερούν οι κυρώσεις τους και τα μέτρα τους. Ω προ αυτό, μπορεί κάποιο από του τρει εμπειρογνώμονε να απαντήσει ξεκάθαρα σε αυτό το ερώτημα. Μην το αποφεύγει το ερώτημα, οι πολιτικοί τα κάνουν αυτά. Η κυρία Σάκε, διαδικαστικό. Βλέπω ότι εκτιμά ιδιαίτερα τους εμπειρογνώμονες ο συνάδελφος. Νομίζω ότι αυτό θα προκύψει και πολλές, σε πολλές άλλες συζητήσεις. Θα ήταν χρήσιμο και σε πολλές άλλες συζητήσεις το σχολείο σας αυτό. Αυτό είπα. Λοιπόν, έχουμε εκπροσώπους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, δημόσιοι πάλι των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Έχετε το λόγο. Ενδεχομένω να πάσχω από Αλτσχάιμερ, αλλά αν θυμάμαι καλά, στην απάντησή μου είπα ότι η βαρύτητα των ΗΠΑ στο χρηματοπιστικό σύστημα δεν μπορεί να παρακαμφθεί και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε και άλλους διάβλους και είπα επίσης ότι το Ιράν χρησιμοποιεί το ευρώ για τις εξαγωγές του. Άρα το ερώτημα είναι τι κάνουμε εμείς. Εμείς προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν το χρηματοπιστωτικό διάβλο ο οποίος είναι πλέον σε ευρώ. Να η απάντηση. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Όχι, όχι, όχι, ολοκληρώνουμε. Ολοκληρώνεται στο σημείο αυτό συζήτηση, λέει ο Πρόεδρο. Και ο Ντέβιτ Μάρτιν, που είναι ο συγητή μα, θα ασχοληθεί με όλα αυτά τα ζητήματα. Ενδεχομένω να άκουσε και κάποιε νέε ιδέε, τι οποίε θα μπορούσε να εντάξει στην έκθεσή του για την αναδιατύπωση. Ο Ντέβιτ Μάρτιν έχει το λόγο. Νομίζω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εξωτερικής Δράσης υπήρξε ειλικρινή μαζί μας ε, ε ως προς ε, τις ενέργειες τις οποίες ε, λαμβάνουμε και πρόκειται για μια δύσκολη διαδικασία την οποία παρόλα αυτά θα πρέπει να ακολουθήσουμε τώρα. Να κάνω κάποια σχόλια πριν περάσω στα συμπεράσματα. Νομίζω πως τα σχόλια που έκανε ο Σάντζο ε, ήταν κάπω ανόητα σήμερα, παρότι τον εκτιμώ ε, γενικότερα, γιατί μα είπε πω ε, συνέκρινε ουσιαστικά την Κίνα με το Ιράν. Η Κίνα είναι ένα με του ισχυρότερου εμπορικού μα τέρου, ενώ με το Ιράν δεν είχαμε εμπορικέ σχέσει για πολύ καιρό. Και μα ρωτάει τώρα γιατί έχουμε και πάλι μια εμπορική συμφωνία. Μα δεν προβαίνουμε σε εμπορική συμφωνία, απλώ έχουμε άρρη τι κυρώσει που είχαμε επιβάλει στο Ιράν. Και Ε, αν θέλει τώρα να μας πει ότι πραγματικά θα πρέπει να μάθουμε πράγματα από ε, τις Ηνωμένες Πολιτείες ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, μια χώρα η οποία μόλις τώρα αποχώρησε από το Συμβούλιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών, από τη Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού και με βάση τα όσα γνωρίζουμε από το ιστορικό των ΗΠΑ σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορούμε να λέμε κάτι τέτοιο. Κάτι ακόμα τώρα προκατακτικά που θα αναφέρω είναι ο, ο, ο συνάδελφος Ντάρμουθ έχει απόλυτο δίκιο ως προς τα προβλήματα ε, του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Πραγματικά αποτελεί αδυναμία αυτό για μας. Ε. Δηλαδή, οι ευρωπαϊκές τράπεζες οι οποίες δραστηριοποιούνται στι ΗΠΑ έχουν περιουσιακά ε, στοιχεία εκεί και πραγματικά αυτό αποτελεί αδυναμία μα αλλά μόνο το τραπεζικό σύστημα θα είναι εκείνο τελικά το οποίο θα ξεφύγει αν θέλετε από τη δική μα προσέγγιση αν ακολουθήσουμε σωστά την προσέγγιση μας στα υπόλοιπα, τομεί. Και αν έχω καταλάβει ε, σωστά, Όπω ισχύει ο Αμερικανικό νόμο, αυτό ε, το, το ΕΝΤΕ επιτρέπει την επιβολή ποινικών κυρώσεων, ε, το οποίο ουσιαστικά αποθανεί και ευρωπαϊκέ επιχειρήσει ότι δηλαδή κάτι τέτοιο μπορεί να αποτελεί ένα πρόβλημα. Πάντως ε, αυτό που θα ήθελα να πω ε, και στον Πρόεδρο είναι ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τις εργασίες μας επί της ε, συμφωνίας με το ΕΡΑ τη Γενικής Συμφωνίας, πράγμα το οποίο αποτελεί και ένα ζήτημα αξιοπιστίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία υπέγραψε αυτή τη συμφωνία, αλλά από εκεί και μετά Νομίζω πως όταν είχαμε προβεί στη διαπραγμάτευση με το Ιράν είχαμε όλοι μας συμφωνήσει ότι θα πρέπει ε, να ακολουθήσουμε αυτή την άγουσα γιατί είναι ο μόνος τρόπος, η προσέγγιση του Ιράν είναι ο μόνος τρόπος ε, όχι επειδή θέλουμε να του συγχωρέσουμε για ό,τι αρέσουν κάνει, απλά επειδή η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν είναι ο ε, μόνο ε, τρόπο ε, για το μέλλον. Και ε, αυτό σημαίνει ταυτόχρονα ότι θέλουμε να επιτρέψουμε στι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει να αναλάβουν πολιτική δραστηριότητα στο Ιράν. Και όπω είπαν και διάφοροι συνάδελφοι, όπω είπε και ο κύριο Αλαφράγκα, το ζητούμενο είναι να βρούμε μια πολιτική ε, συμφωνία έτσι ώστε να μην έχουμε και εξωεδαφικές συνέπειε από άλλες ε, ε, ε, διατάξεις. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια θα λειτουργήσουν και τέτοιου είδους κυρώσεις, αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον και από εκεί και μετά θα πρέπει να διασφαλίσουμε την προστασία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν κυρώσει και ήδη εργάζεται από αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί πραγματικά κάτι τέτοιο είναι πολύ αρνητικό ως επίπτωση. Ε, γιατί ακόμα κι αν εμείς ε, προβλέψουμε αυτές τις διατάξεις, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορεί να αποσυρθούν από την αγορά του Ιράν μόνο και μόνο επειδή φοβούνται ότι ενδεχομένως μπορεί να προκύψει ε, να υπάρξει μια απειλή για αυτές στο μέλλον. Οπότε καλό είναι το ότι προετοιμάζει κάποια μέτρα η Επιτροπή, αλλά περισσότερο ε, μακροπρόθεσμα, όχι τώρα άμεσα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει μία αναθεώρηση του βασικού κανονισμού. Αλλά αντιλαμβάνω βέβαια ότι προς το παρόν λόγο και του επίγοντος χαρακτήρα του ζητήματο θα πρέπει να προβούμε εδώ σε ένα εργαστήριο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο, για αυτέ τι σαφεί συμβουλέ και συστάσει που μα δώσατε σε ό,τι αφορά τι μελλοντικέ εργασίε και θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε αυτό το ζήτημα και μετά από το καλοκαιρινό μα διάλειμμα. Ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Οπότε θα διακόψουμε τώρα για λίγο και μετά από αυτό το σύντομο διάλειμμα θα συνεχίσουμε με τη συνεδρίαση των συντονιστών. Συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών, οπότε, οπότε όσοι δεν επιτρέπονται δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν σε αυτή την συνεδρίαση των συντονιστών θα πρέπει να αποχωρήσουν από την αίθουσα. Και ίσως οι πολιτικές ομάδες θα μπορούσαν να ζητήσουν από τους συντονιστές τους να προσέλθουν στην αίθουσα λίγο νωρίτερα.